Ακόμη και αν πολλοί συνάδελφοι δεν σεβάστηκαν την πρόσκλησή μου για απόλυτη συνέπεια στις 3 και 4 πρέπει να βιαστούμε να ξεκινήσουμε γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας για το απόγευμα. Ξεκινάω λοιπόν τη συνεδρίαση με το πέμπτο σημείο στην ημερήσια διάταξη που αφορά στην παρουσίαση μίας μελέτης που η Επιτροπή μας ζήτησε πώς να δημιουργήσουμε ένα διακρατικό κομματικό σύστημα. Ένας από τους συγγραφείς, ο, Λουτσάνο, ο καθηγητής Λουτσάνο Μπάρντι που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό ε, Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, είναι εδώ και θα τον παρακαλέσουμε να μας παρουσιάσει μία περίληψη της εργασίας αυτής και in extenso το κείμενο θα το βρείτε στα έγγραφά σας. Είστε εδώ από το πρωί, ακούσατε τι είπαμε λίγο πολύ και θα μας διαφωτίσετε ακόμη περισσότερο πώς λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα διακρατικό κομματικό σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πάω αμέσως στα αγγλικά, γιατί η παρουσίαση είναι στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Πολλά μέλη της Επιτροπής ήδη έχουν λάβει μια προκαταρκτική πρωτόλια έκδοση της έκθεσης. Θα ήθελα να τονίσω περισσότερο τη μέθοδο που χρησιμοποίησαμε στα, στη μελέτη μας και να καταλήξω σε ορισμένα συμπεράσματα και πορίσματα αυτής της μελέτης. Το σχέδιο που ήταν η βάση της έκθεσης ήταν το γεγονός ότι το Νοέμβριο του 2009 το Παρατηρητήριο Πολιτικών κομμάτων και εκπροσώπηση ε, κέρδισε ένα διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, προκειμένου να καταρτήσει μια μελέτη για την ανάπτυξη ενό ε, διακρατικού συστήματος κομμάτων. Έτσι δημοσιεύθηκε η έκθεση που αναλύει τον αντίκτυπο της ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός συστήματος διακρατικών κομμάτων. Απαρτίζεται από τέσσερα σημεία η μελέτη και κάθε ένα από αυτά αφορά σημαντικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού συστήματος. Ομογένεια, η ε, μεγάλο μέγεθος, η πρακτική επιλογή υποψηφίων, πολιτική παιδεία και οργάνωση του κόμματος, σύγκληση σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση του κόμματος και εκλογική νόμη. Το πρώτο τμήμα αφορά την ομοιομορφία, την ομογένεια στην ιδεολογική τοποθέτηση. Και μάλιστα η διαφάνεια αυτή σχετίζεται με την επόμενη που περιλαμβάνει κάποια, κάποιους πίνακες ιδεολογικής τοποθέτησης των εθνικών κομμάτων και πώς ε, αντα, αντανακλώνται αυτά στην ευρωπαϊκή, σε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Εδώ έχουμε τρεις ε, τέτοιες, ε, τρία τέτοια σχήματα. Έχουμε την ευημερία, των τον α, ε, φιλελεύθερο σοσιαλισμό, τις οικονομικές ελευθερίες, τα οικονομικά ζητήματα, νομιμότητα, μετανάστευση και περιβάλλον. Αυτές είναι οι διαστάσεις που φέρονται σε αυτό το ραχνοειδές διάγραμμα και με βάση έρευνες που κάναμε και δημοσκοπήσεις βλέπουμε τη θέση των εθνικών κομμάτων και των ομάδων κομμάτων. Υπάρχει, βλέπετε, ένας επαρκής βαθμός ομοιομορφίας, ομοιογένειας μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεγαλύτερη ομοιογένεια παρατηρείται στους φιλελεύθερους. Ενώ υπάρχει λιγότερη ομοιομορφία, ομοιογένεια στις άλλες τρεις ομάδες. Και φυσικά υπάρχει μια πιο αριστερή τάση στην ε, Ενωμένη Αριστερά και στους Πρασίνους. Βέβαια, στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής επικράτειας χρειαζόμαστε ομοιόμορφες, ομοιογενείς πολιτικές ομάδες. Και αυτό αφορά και τις προγραμματικές τους δηλώσεις και την ιδεολογική τους θέση. Θέλουμε δηλαδή οι εκλογές οι ψηφοφόροι που συνήθω έχουν σημείο αναφορά τα κόμματα σε εθνικό επίπεδο, να μπορούν να ταυτίζονται και να αισθάνονται άνετα με τα προγράμματα που θα παρατηρούν τα προεκλογικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε η απέτηση πολιτική συνάφεια μεταξύ κάποιων ομάδων είναι σημαντική προϋπόθεση, όχι μοναδική μόνο, για τέτοια πολιτική τοποθέτηση και τη διαμόρφωση μιας πολιτικής κουλτούρας. Τώρα, η μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, που ήταν η διεύρυνση για τη συνοχή των πολιτικών ομάδων, είχε περιορισμένη εμβέλεια ή τουλάχιστον είχε πιο περιορισμένη από ό,τι περιμέναμε. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε με θετική σκοπιά. Και φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα της ε, ομοιομορφίας των ομάδων, γιατί έδειξαν οι έρευνες ότι διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και την ομοιομορφία, ομοιογένεια των πολιτικών ομάδων. Επίσης θα πρέπει να είναι εμφανείς οι ιδεολογικές τοποθετήσεις ε, και η διάκριση μεταξύ πολιτικών αριστεράς και δεξιάς. Μπορείτε να εξετάσετε αυτά τα γραφήματα και πιο εκτεταμένα μπορώ να σας μοιράσω αυτούς τους πίνακες, αυτούς που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Προχωράμε στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης που πραγματεύεται τις πρακτικές της επιλογής υποψηφίων. Η έλλειψη ομοιομορφίας στην ε, επιλογή υποψηφίων εντό των πολιτικών ε, ευρωπαϊκών οικογενειών μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσκομα σε, μια, σε ένα πραγματικά διεθνικό διακρατικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών κομμάτων. Και αυτό είναι το πόρισμα, το αποτέλεσμα των παρατηρήσεών μας, που πιο διεξοδικά φυσικά αναλύονται στην έκθεση. Οπότε αυτά τα πορίσματα που σας παρουσιάζω τώρα είναι αυτό που βρήκαμε μετά από τη διεξοδική ανάλυση που κάναμε. Δεν είναι αξιώματα αυτά που σας παραθέτω, είναι ο καρπός μιας διαδικασίας ανάλυσης. Όσο είναι μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα της επιλογής, τόσο μπορούν ψηφοφόροι να ψηφίζουν περισσότερο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομάδα παρά την Εθνική, το Εθνικό Κόμμα. Αυτό μπορεί να φαίνεται, φαίνεται ως παράδοξο, αλλά από άποψη αποκέντρωσης ήταν ένα πόρισμα της έκθεσης. Και η πιο συνηθισμένη διαδικασία αφορά το ρόλο του εκτελεστικού Συμβουλίου των Κομμάτων και του Συνεδρίου των Κομμάτων. Σε με το 86% από όλες τις προτάσεις που προκύπτουν από το εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η περιγραφή μιας κατάστασης που ίσως θα ζητήσουμε να τροποποιηθεί κάπως. Το τρίτο τμήμα της έκθεσης αφορά τις πολιτικές κουλτούρες και την οργάνωση. Η μεγάλη ποικιλομορφία των κομμάτων σε εθνικό επίπεδο και η παρουσία δύο περισσότερων εθνικών κομμάτων μέσα σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Κομματικού Συστήματος. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κατακαιρματισμός σε εθνικό επίπεδο των συνιστοσών μιας συγκεκριμένη ε, ομάδα κομμάτων και η ταυτόχρονη παρουσία δύο ή περισσότερων κομμάτων από την ίδια χώρα ενός ε, εντός μιας συγκεκριμένης ομάδας κομμάτων μπορεί να δημιουργήσει τριβές και εντάσεις, ακόμη και στην εξέλιξη μιας ε, ομάδας κοινοβουλευτικής. Γιατί μπορεί να προσδιορίζεται από εθνικά στοιχεία περισσότερο και εθνικές αντιπαραθέσεις. Ο κίνδυνος λοιπόν έγκυται στο εξής. Πώς θα καταφέρουμε να μεταφέρουμε από από να μην, να μην ε, μεταφέρουμε από το εθνικό επίπεδο κάποιες αντιζηλείς αντιπαλότητες από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές κουλτούρες πάντως και την οργάνωση, το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κόμματα υπόκειται στο ίδιο νομικό καθεστώς ε, ή ίσως μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ε, Ευρωπαϊκού Συστήματος Κομμάτων. Και μάλιστα το πρωί ασχοληθήκατε με τα θέματα αυτά και για τα θέματα αυτά θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα όταν θα μου ξαναδώσετε το λόγο. Η, η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος α, εξαρτάται και από τις πολιτικές κουλτούρες και από τον τρόπο επιλογής. Να είναι γνωστό αυτό το σύνδρομο και η σημασία που αποδίδεται ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο στις ευρωεκλογέ είναι πραγματικά ε, η αξία συλληδία λιδίας λίθου. Και μάλιστα όχι μόνο για πολιτικά ζητήματα και όχι μόνο για πολιτικά θέματα που ενδιαφέρουν σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για τις ε, στρατηγικές των κομμάτων. Γιατί τα κόμματα δοκιμάζουν κατά κάποιο τρόπο ορισμένους οργανωτικούς τους στόχους στις ευρωεκλογές πρώτα. Τις ευρωεκλογές τη χρησιμοποιούν ως λιθο. Και αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα σε ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές ομάδες ή κόμματα. Η χρηματοδότηση των κομμάτων τώρα και η εκλογική νόμη, ένα θέμα που αναλύσατε το πρωί. Το αναφέρουμε και στην έκθεση, αλλά με κάπως διαφορετικό τρόπο. Αυτά που είπατε το πρωί θα τα σχολιάσω αργότερα. Εγώ θα σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα της έκθεσης που όπως σας είπα δημοσιεύθηκε πριν από μήνες. Φυσικά, πρώτα ασχοληθήκαμε με τους εκλογικούς νόμους. Η προτινόμενη διακρατική εκλογική περιφέρεια μπορεί να ενισχύσει την, την στενότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας πραγματική διακρατική προεκλογική εκστρατεία και ευρωπαϊκά ή πανευρωπαϊκά προεκλογικά προγράμματα. Νομίζω ότι αυτή είναι και κρατούσα γνώμη προς αυτό. Σε ό,τι αφορά την ε, προτιμησιακή ψήφο που όταν εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να έχει ε, θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα αν καταφέρουμε να δείξουμε στους ψηφοφόρους ότι η έρευνα έχει αποδείξει ότι η προτιμησιακή ψήφος είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία και μέσα που έχουν οι ψηφοφόροι στη διάθεσή τους για να επηρεάσουν την... τους βουλευτές, την συμμετοχή των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, που εξαρτώνται συνήθως από τις ε, επιλογές, τις κομματικές επιλογές. Αν υπάρχει όμως ε, πραγματική και ψήφος, ψήφος προτίμησης μάλλον, έχουμε την άμεση ε, επέμβαση ουσιαστικά του ψηφοφόρου. Και ουσιαστικά η προεκλογική συμπεριφορά μπορεί να καθορίσει το κατά πόσο θα επιλεγεί ο συγκεκριμένος ε, ευρωβουλευτής. Ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα κομματικής χρηματοδότησης μπορεί να προωθήσει μια σύγκληση οργανωτική. Και αυτό το πόρισμα στηρίχθηκε σε μια σειρά παρατηρήσεων που αναλύονται στην έκθεση και παρουσιάζονται πιο διεξοδικά. Παρά τα θετικά κίνητρα που δίνονται από, που δόθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2004-2003, τα πολιτικά κόμματα ευρωπαϊκού επίπεδου υπόκεινται ουσιαστικά στις εθνικές συνιστώσεις και τα, τις ε, κοινοβουλευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα τα διεθνικά κόμματα ή διακρατικά κόμματα έναντι του διεθνικού κομματικού συστήματος. Η θέση μας, και νομίζω ότι κάποιος είπε το ίδιο και το πρωί, ότι το κομματικό σύστημα δεν απαρτίζεται από το άθροισμα των κομμάτων, αλλά και από τις ε, ε, αλληλεπιδράσεις τους και τους περιορισμούς που υφίστανται τα κόμματα. Δηλαδή, τα κόμματα προηγούνται του κομματικού συστήματος. Αυτή τουλάχιστον ήταν η δική μας εμπειρία ε, στις νέες δημοκρατίες, στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Και πιστεύουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο όπου πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο σύστημα των διακρατικών κομμάτων, αλλά δεν έχουμε ακόμη ένα διακρατικό κομματικό σύστημα. Για παράδειγμα, σε εθνικό επίπεδο έχουμε το, το βελγικό σύστημα, αλλά μπορεί να έχουμε ακόμη και δύο κομματικά συστήματα στο Βέλγιο. Αλλά δεν έχουμε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο κομματικό σύστημα. Τώρα, ως προς τα κίνητρα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα, ενάυσματα, για να προωθηθεί η πολιτική αλληλεπίδραση μεταξύ των κομμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα πορίσματα, τα συμπεράσματα της έκθεσης και ίσως και κάποιες συνταγές που θα προτείνουμε. Η ανάπτυξη διακρατικών κομμάτων είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός διακρατικού κομματικού συστήματος. Το βασικό πρόβλημα έγκαιται στην έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των κομμάτων για τον έλεγχο των εκτελεστικών σωμάτων. Αυτό αναφέρθηκε και το πρωί και επιμένουμε και εμείς αυτό. Δεδομένου του θεσμικού πλαισίου, ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να αυξηθεί, να ενισχυθεί μέσω συντονισμού των κοινοβουλευτικών απαντήσεων στις νέες ε, διαδικασίες ό,τι αφορά τις παραβιάσεις ε, της αρχής της επικουρικότητας και προτείνοντας υποστήριξη του δικού τους, των δικών τους υποψηφίων για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θα πρέπει να γίνει τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Να διευρύνουμε τους ε, κομματικούς δεσμούς ε, σε, σε επίπεδο βάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, να εξετάσουμε τα κόμματα την ομάδα μας ως ε, σύνολα τριών οργανωτικών ε, συστατικών της βάσης, του, των κομματικών γραφείων και του κεντρικού γραφείου. Και το κεντρικό γραφείο είναι οι παλιές ομοσπονδίες. Τώρα, να δημιουργήσουμε έναν ε, πανευρωπαϊκό κομματικό ανταγωνισμό, να προωθήσουμε την προβολή των κομμάτων και την ευρωπαϊκή τους διάσταση και ανάλογα με το πώς θα γίνουν όλα αυτά, θα σας το πω σε μια ώρα που θα ξαναλάβω το λόγο για μια δεύτερη παρουσίαση. Ευχαριστώ. Bene, professor Bardi, la ringraziamo. Σας ευχαριστούμε καθηγητά Μπάρντι. Εσείς ε, ήδη στη φάση της επεξεργασίας ε, του σχεδίου μας είχατε δώσει μια avant première, είναι έτοιμο, μπορούμε να το διαβάσουμε. Όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις ή τοποθετήσεις, Γκερέρο. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά Μπάρδη για την παρουσίασή σας. Δυστυχώς χάθηκα στο πρώτο τμήμα της παρουσίασης και θα ήθελα να εκφράσω μία σκέψη για ένα τμήμα που το θεωρώ σημαντικό διότι δεσμεύει αυτή την μελέτη για τα συστήματα ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων με μία ε, εκλογική μεταρρύθμιση, που, ε, μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος που συζητάμε εδώ ε, στην Επιτροπή και που αφορά στην προτιμησιακή ψήφο. Η προτιμησιακή ψήφος συνδέεται με την ποιότητα της ε, δημοκρατίας υπό την έννοια ότι ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να εκτιμήσει την πρόταση που του, κάνει, του υποβάλλει ένα κόμμα, αλλά να επηρεάσει εκλέγοντας αυτόν που προτιμάει. Αυτό δηλαδή είναι ένα μέσο κατά της γραφειοκρατίας ή του, του υπερβολικού συγκεντρωτισμού των κομμάτων. Όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι ανάλογα με την πολιτική κουλτούρα των κρατών λειτουργεί είτε προς τη μία κατεύθυνση αλλά μπορεί να λειτουργήσει και προς την άλλη. Δηλαδή η προτιμησιακή ψήφος στην στη Γερμανία κανένας δεν την αμφισβήτησε. Ενώ όμως στην Ιταλία, ναι, κυρίως στην Νότιο Ιταλία. Και αυτό στο βαθμό ότι η προτιμησιακή ψήφος μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικές εκστρατείες, σε μεμονωμένη χρηματοδότηση υποψηφίων είτε και ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων του ιδίου κόμματος. Αυτό σε εθνικό επίπεδο. Τώρα εμένα η αμφιβολία μου για το προτιμησιακό σύστημα ε, μέσα στο σύστημα της διακλατικής ψηφοφορίας διεθνικής ψηφοφορίας. Είτε θα γίνεται έτσι όπως, άμα, όπως γίνεται σήμερα, θα οδηγούσε αυτούς που έχουν περισσότερο πληθυσμό να εκλέξουν τους δικούς τους υποψηφίους με τη δική τους εθνική προέλευση. Δηλαδή αν για, για μια λίστα 25 ατόμων οι Γερμανοί ψηφίσουν τον Γερμανό ή οι Ισπανοί τον Ισπανό, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε 46 εκατομμύρια ή οι Ιταλοί τον Ιταλό, οι δυνατότητες εκλογής του Λιθουανού, του Μαλτέζου ή οποιοδήποτε άλλου θα μειωνόντουσαν αισθητά. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διαφορετική υπόθεση μπροστά μας ότι η διαπραγμάτευση της σύνθεση του ψηφοδελτίου θα είναι μία διαπραγμάτευση μεταξύ κομμάτων οι πολίτες θα αποφάσιζαν αλλά θα έχουμε ένα ψηφοδέλτιο πάνω από 25 άτομα και θα αποφασίζουν οι πολίτες Τώρα αυτή είναι μια πρώτη σκέψη σε μια δεύτερη φάση όπου θα έχουμε ένα θεσμοθετημένο σύστημα κομμάτων και ένα εκλογικό σώμα με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνείδηση και πιο διαχειμένη εθνική συνείδηση θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να ρωτήσει. Παρακαλώ λοιπόν τον καθηγητό Μπάρτι να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Γκερέρο. Βεβαίω. Επειδή μιλάμε για προτιμησιακή ψήφο θα, μιλήσουμε, θα μιλήσουμε ιταλικά. Λοιπόν, συμμερίζομαι όλα τα σημεία που ανέφερε ο κύριος Γκερέρο να διευκρινίσω όμως μερικά πράγματα τεχνικού χαρακτήρα. Διότι η συντομία της προηγούμενης μου παρουσίασης δεν μου επέτρεψε να εξηγήσω όταν εμείς μιλούσαμε για προτιμησιακή ψήφο ε, υποβάλαμε μία τεχνικού χαρακτήρα συμβουλή την πολιτική λύση την ε, βρει, θα την βρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι δική μας δουλειά. Και αυτό, αυτή την πρόταση θα την υποβάλαμε μέσα από, όταν θα είχαμε έναν νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος θα εφαρμιζόταν σε όλους τους βουλευτές και όχι μόνο στην διεθνική εκλογική περιφέρεια. Και αυτό γιατί φοβηθήκαμε ότι οι μικρότερες χώρες θα είχαν το πρόβλημα όπως εσείς το αναφέρατε. Για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη χρήση που μπορούμε να κάνουμε πάλι από τεχνικής πλευράς. Εγώ νομίζω ότι μέγα μέρος των προβλημάτων που συνδέονται με την προτιμησιακή ψήφο και την κακή χρήση που γινόταν και συνεχίζει η μέρη να γίνεται ακόμη στην Ιταλία, αυτό έχει να κάνει με τις πολλαπλές επιλογές. Άμα είχαμε μόνο ένα σταυρό για έναν υποψήφιο, μέγα μέρος αυτών των προβλημάτων αποφεύγονται. Σίγουρα είναι πρόωρο ε, το θέμα. Μπορώ να το δεχτώ. Αλλά την πρώτη μελέτη που έκανα εγώ για το, για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκανα το 1987, πέρασαν σχεδόν 24 χρόνια. Και τότε ήταν πρόορη η λύση όταν ε, μεταρρυθμίστηκε το Βρετανικό εκλογικό σύστημα η λύση θεωρήθηκε πρόορη ε και πάλι πρόορη είναι, ανώριμη είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων εγώ εδώ είμαι και όποτε μου το ζητάτε σας δίνω τη γνώμη μου. Κύριος Βίλαντ. Συγγνώμη που ζητώ μετά το λόγο, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι πολύ περισσότεροι θα δηλώνονταν. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Νομίζω ότι για την συζήτησή μας θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας τι καινοτομίε μπορούμε να εισαγάγουμε βραχυπρόθεσμα. Γιατί κάποιες προτάσεις σας προϋποθέτουν εφαρμογή μέσα από τροποποίηση του πρωτογενούς δικαίου. Άλλες προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν μέσω του δευτερογενούς δικαίου και άλλα είναι πολιτικές ε, απαιτήσεις. Ας πούμε, οι οικογένειες των κομμάτων που έχουν συνοχή θα πρέπει να ε, αποφασίζουν και για έναν ε, κοινό πολιτικό υποψήφιο. Αυτό είναι θέμα πολιτικής εφαρμογής. Όταν μιλάμε λοιπόν για ε, συγκρότηση κομμάτων σε διεθνικό επίπεδο, πάντα νιώθω ότι κάτι λείπει, γιατί πολλά συνεπάγονται ε, τροποποίηση της συνθήκης ε, από πού θα προέρχονται οι υποψήφοι, από πόσα κράτη, κάποια κράτη-μέλη μπορούν να διαφοροποιηθούν ή να διαφωνήσουν και να ζητήσουν πιο ισορροπημένη λύση για να μην δοθούν σε ορισμένους ε, υπερβολικά προνόμια. Πριν από το 2019 θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να γίνει. Πιο σημαντικό είναι και πιστεύω ότι με το, την εξέλιξη του κανονισμού των κομμάτων είναι το θέμα της εσωκομματικής δημοκρατίας. Αυτό το θέμα νομίζω ότι είναι σημαντικό εφόσον θα συζητήσουμε την νομιμοποίηση των εκλογών και της εκλογής του υποψηφίου και πόσο νομότυπη και πόσο νομιμοποιείται ε, μία προβολή υποψηφίου. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να συνδέσω με κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως ορισμός υποψηφίων με μυστική ψηφοφορία και ελάχιστα πρότυπα επαρκή, εις ό,τι αφορά την συμμετοχή στις εκλογές σε εθνικό επίπεδο. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να ακούσω περισσότερα πράγματα. Η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Έχει πολύ ενδιαφέρον η έρευνα που έγινε κατόπιν εντολής της δικής μας Επιτροπής ε, γιατί μπαίνει σε μεγαλύτερο βάθος όπως έχετε σημειώσει το να δημιουργήσει κανείς πανευρωπαϊκά κόμματα δεν σημαίνει ότι δημιούργησε αυτομάτως και ένα σύστημα ευρωπαϊκών κομμάτων. Και αυτό είναι ευθέως αντιληπτό. Βεβαίως, η εξέλιξη ορισμένων ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε γίνεται βήμα προς βήμα. Θα μπορούσα να πω ότι βλέπει κανείς σήμερα κάτι να συζητιέται, αύριο διατυπώνεται σε ένα χαρτί και μεθαύριο το βλέπει με έκπληξή του να αρχίσει να πραγματοποιείται. Δεν μπορεί βεβαίως να μιλήσουμε για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής λίστας κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές αν δεν έχουμε ένα σύστημα ευρωπαϊκών κομμάτων. Ένα σύστημα που να υπακούει σε ένα κοινό στάτους και που να έχει βέβαια αυτό που αναφέρετε εσείς και είναι πολύ σωστό τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών κομμάτων. Επομένως αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, γιατί η έκθεση είναι βέβαια για τη χρηματοδότηση, είναι να γίνει ουσιαστικά το πρώτο βήμα, δηλαδή να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ε, βάσει ενός κανονισμού που θα έρθει ως πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις ελάχιστες αλλά αναγκαίες προϋποθέσεις πρώτον για τη δημοκρατικότητα αυτών των πανευρωπαϊκών κομμάτων και για τις σωστές επιλογές περαιτέρω αυτό που εγώ ήθελα να σας ρωτήσω είναι, επειδή ετέθη το πρωί, πώς βλέπετε τη δυνατότητα αυτών των κομμάτων να μην εντάσσουν μόνο κόμματα μέλη από τις διάφορες χώρες, αλλά να εντάσσουν ταυτόχρονα και έναν οποιοδήποτε αριθμό, όσο μεγάλος και αν είναι, φυσικών προσώπων από τα κράτη-μέλη που δεν επιθυμούν να ενταχθούν κατά ανάγκη στα εθνικά τους κόμματα ή και φυσικών προσώπων που προέρχονται από χώρες που δεν υπάρχουν κόμματα μέλη σε ένα κόμμα αυτού του χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την παρατήρηση του κυρίου Βίλαντ Μα νομίζω ότι απευθυνόντουσαν περισσότερο στον κύριο Γκερέρο και όχι σε μένα. Ε, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν συνταγματικές πλευρές ε, πρωτογενές και δευτερογενές δίκιο πέρα από τα πολιτικά δηλαδή και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο λύσεις από μένα που έρχομαι εδώ ως εμπειρογνώμονας και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να, εκφράσω τι θα ήταν ευκταίο. Η σύστασή μας λοιπόν για το κατά πόσο θα πρέπει να προταθεί ένας υποψήφιος των κομμάτων για, την Κομισιόν. Ε, αυτό το εξαρτάται από τα κόμματα. Και ορισμένα από αυτά τα κόμματα έχουν αυτόν τον προσανατολισμό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να δώσει ε, ένα έναυσμα για, την, ε, για τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ε, μπορέσει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός, ενός συστήματος. Αυτά για τις παρατηρήσεις της εισηγήτριας. Τώρα, για τη συνταγματική μεταρρύθμιση που θα χρειαζόταν ή στο πρωτογενές δίκαιο για τον ορισμό της ε, διεθνικής εκλογικής περιφέρειας Μα αυτό θα το αποφασίσει αυτή η Επιτροπή. Εμείς θεωρούμε ότι αν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αν ήταν εφικτό θα ήταν ευκταίο. Η ψήφος εμπιστοσύνης, η προτιμησιακή συγγνώμη ψήφος, όπως υπόθηκε, για ορισμένους όρους, υπό όρους μπορεί να εγκριθεί. Και είναι ευκταίο και το θέμα των διορισμών που ανέφερε ο κύριος Βίλαντ για το θέμα του ανήκειν, του membership των πολιτών που μπορεί να μην είναι μέλη των εθνικών κομμάτων. Θα, το, θα μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Εμείς στην ερευνητική ομάδα που εκπροσωπώ συμφωνούμε αλλά όχι με μία, απαραίτητα με μία παραδοσιακή μορφή μέλους κόμματος διότι αυτού του είδους το πολιτικό ανήκει βρίσκεται σε παρακμή και σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή οι supporters, τα μέλη των κομμάτων και των επισήμων μελών είναι ευκαιρία αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια άλλου είδους μορφή ε, κομματικού ανήκειν διαφορετική από αυτή των εθνικών κομμάτων. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι άσπρα μαύρα, υπάρχουν πάντοτε ε, πολλά στοιχεία που μπορούμε να βρούμε για την υπέρ της μίας ή της άλλης λύσης. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε όμως είναι η αλλης λυσης εμεις αυτο το σπουδειο θελουμε τέλο πάντων το, το ανήκει σε ένα κόμμα, να μην βρίσκεται σε αντίφαση με το Εθνικό Κόμμα. Ο κύριος Γερερό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω στον ε, κύριο Βίλαντ ότι εγώ απλώς αναφέρθηκα στην έκθεση του Άντριου Νταφ για την εκλογική μεταρρύθμιση και το βασικό περιεχόμενο σήμερα είναι να δημιουργηθεί ένα, διεθνικό ψηφοδέλτιο 25 ε, υποψηφίων. Δεν είναι ότι δεν το πρότεινα εγώ, ο Άντριου Ντάφ το πρότεινε. και για για το να παρουσιαστεί ένας υποψήφιος από τα ευρωπαϊκά κόμματα και να υποδειχθεί ως επίτροπος σε η πρόεδρος της Κομισιόν άμα κερδίσει το κόμμα της εκλογές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, μπορεί να ψηφίζουν ευρωπαϊκά οι πολίτες στις ευρωεκλογέ και να χρησιμοποιήσετε όλα τα επιχειρήματα. Αλλά όταν πάνε στην κάλπη παρά το πολιτικό επιχείρημα ε, είναι, ε, αντιδρούν αυτόματα σαν να ψηφίζουν το Εθνικό Κόμμα για την Εθνική Κυβέρνηση. Στις περιφερειακές εκλογές στην Ισπανία η συμμετοχή κατεβαίνει στο 60% και στις ευρωεκλογές κατεβαίνει στο 45% και 70% όταν συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές. Έχουμε 30 πόντους όμως διαφορά. Και όταν πολλούς πολίτες τους ρωτάμε, σε μεγάλο βαθμό μας λένε ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν όταν ψηφίζουν για τις ευρωεκλογέ. Ξέρουν όμως πάρα πολύ καλά ότι εκλέγουν κυβέρνηση όταν ψηφίζουν στις γενικές εκλογές. Οπότε, ότι μπορεί να οδηγήσει προς μία αποφασιστική εκλογή, δηλαδή ο ψηφοφόρος έχει συνειδητοποιήσει ότι αποφασίζει για κάτι, κάτι σοβαρό που έχει να κάνει με την διακυβέρνηση και το, το δικό του πολιτικό προσανατολισμό, αυτό είναι καλό και για την πολιτική του συμμετοχή. Και το Ευρωπαϊκό Κομμουνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα εκτιμά αυτή τη δυνατότητα να κατεβάσει ε, έναν υποψήφιο πρόεδρο για την Κομισιόν στις εκλογές του 2014. Πρόκειται για κάτι το οποίο de facto έγινε στο παρελθόν στις προηγούμενες εκλογές ακόμη και χωρίς να είναι δηλαδή εντελώς καθαρό υπήρχε μία συνείδηση ότι το ΕΛΚ παρουσίαζε ως υποψήφιο τον κύριο Μπαρόσο. Δεν υπήρχε βέβαια ένα σαφές πολιτικό μήνυμα στην κατά την προεκλογική εκστρατεία. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει κάτι τέτοιο το 2014. Αν δηλαδή ο πολίτης, ε, και έτσι μάλλον ο πολίτης μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αποφασίζει για κάτι πιο συγκεκριμένο και πιο απτό και σοβαρό. Ή ο κύριος Χέφνερ. Αλλά ξανά, πρόταση που έκανα εγώ το πρωί. Προβλέφθηκε στο πρόγραμμα ότι από τις 4 ως τις 5 πρέπει να ακολουθήσουμε, να ακούσουμε εδώ τους τέσσερις καθηγητές και μετά ξανά τον καθηγητή Μπάρντι. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε τη γενική συζήτηση μετά τους ομιλητές. Μπορώ να περιμένω, λέει ο κύριος Ράντζα. Ωραία, τότε να προχωρήσουμε. Παρακαλώ λοιπόν τον καθηγητή Μόρλοκ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Γερμανικό Ίδρυμα για τα πολιτικά κόμματα. Ένα τέταρτο έχει στη διάθεση, έχουν στη διάθεσή τους οι τέσσερις εμπειρογνώμονες για σήμερα. Ο, ο καθηγητής Μόρλοκ, ο καθηγητής Μπάρν, α τρεις είναι οι καθηγητές, Α, και είναι και ο καθηγητής Χρυσοχώμα, να προφέρω καλά τα ελληνικά, δεν ξέρω τι λέτε. Λοιπόν, ο καθηγητής Μόρλοκ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, δημοκρατία τι σημαίνει δυνατότητα επιρροής της πολιτικής εξουσίας. Καλή δημοκρατική τάξη ε, δημιουργεί διάβλους ώστε όλα αυτά να ε, γίνονται. Αυτά τα θεσμοθετημένα κανάλια ή διάβλους εισρωής είναι η διαβλους ροης ειναι η κριτικη ε, ε, κοινή γνώμη, τα κόμματα και άλλοι μηχανισμοί άσκησης επιρροής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οι ειδικοί οργανισμοί, τα πολιτικά κόμματα τι είναι. Είναι ειδικοί οργανισμοί, οργανώσεις για την άσκηση πολιτικής επιρροής. Μπορούμε να το δούμε και αντίστροφα. Η πολιτική επιρροή διευκολύνεται πολύ περισσότερο ή στο βαθμό που υπάρχει καλά εδρεωμένο κομματικό σύστημα. Η καλή δημοκρατία, αν θέλετε, προϋποθέτει λοιπόν κόμματα σύστημα των κομμάτων. Αυτή είναι μια βάση που μας βρίσκει όλους σύμφωνους ως σημείο εκκινήσεως. Διαπιστώνουμε όμως ότι στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα υπάρχουν πολιτικές επιρροές που περιορισμένα ε, περνούν από τα πολιτικά κόμματα και ακόμα πιο ε, περιορισμένα από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα γιατί οι βασικοί ε, είναι οι εθνικές κυβερνήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια, ε, και κόμματα. Βεβαίως, εδώ δεν ξεχνάω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σωστό ότι το άρθρο 10 της ε, συνθήκης της Ένωσης που αναφέρεται στη Δημοκρατία, στην παράγραφο 4, ξανά αναδεικνύει το ρόλο των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν δρούν μόνο στο κοινοβούλιο, αλλά τα πολιτικά συμφέροντα, οι πολιτικές συγκρούσεις σε όλο, σε όλο τους το εύρος ε, λαμβάνονται υπόψη από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Άρα είναι κεντρικό καθήκον να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα κομματικών, ένα σύστημα ευρωπαϊκών κομμάτων. Συμφωνώ εδώ με τον συνάδελφο Μπάρντι. Γνωρίζουμε, όπως είπαμε και όλας, ότι μέχρι τώρα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν περιορισμένη σημασία. Οι, ευρωπαϊκές, οι ευρωεκλογές επηρεάζονται από εθνικά θέματα. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να αναζωογονήσουμε το ε, σύστημα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Τρία σημεία θα αναφέρω εδώ. Πρώτον, το θεσμικό πλαίσιο, πρώτον, τα δημοσιονομικά δεύτερον και οι ε, κομματικοί κανόνες, κανονισμοί ε, σε ειδικότερο επίπεδο. Το πρώτο θέμα είναι πολύ σημαντικό γιατί τα κόμματα αναπτύσσονται σωστά στο βαθμό που υπάρχουν ε, και τομείς ανάληψης δραστηριοτήτων για τα κόμματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κοινοβουλευτικό πλαίσιο το οποίο θα τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται. Εδώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκού επίπεδου και εθνικού επίπεδου. Και ε, πρέπει να σκεφτούμε εδώ το ρόλο που, παίζουν, που παίζει η συνθήκη. Τι τομείς δραστηριοτήτων μπορεί να ενδιαφέρουν και να προσελκύουν τα ε, κόμματα. Και θα πρέπει να δούμε μήπως μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς τους τομείς ανάληψης δραστηριότητας για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Θα επανέλθω σε αυτό. Δεύτερον, τα χρήματα. Χρήματα χρειάζονται για τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να μην εξαιρέσουμε εδώ και την ανάγκη για χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και από τον προϋπολογισμό που θα επιτρέψει καλύτερη λειτουργικότητα στα κόμματα. Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό μπορεί να είναι ένας μηχανισμός ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των κομμάτων και βεβαίως αυτό επηρεάζει και την πολιτική ισότητα ευκαιριών. Ε, τα κόμματα καλύπτουν και αντανακλούν διαφορετικά φάσματα και τομείς της κοινωνίας και ε, ορισμένα μπορεί να προβάλλονται περισσότερα από άλλα. Γι' αυτό η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δημιουργεί μια εξίσωση στην αντιμετώπιση των κομμάτων ή τουλάχιστον συμβάλλει σε αυτήν. Το τρίτο θέμα που θα με απασχολήσει είναι η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού στάτους των κομμάτων και του κανονισμού των ευρωπαϊκών κομμάτων. Υπάρχουν δέκα ερωτήσεις από την πλευρά σας και βασίζομαι σε αυτές. Καταρχήν το θέμα της, ε, του νομικού προσώπου. Πράγματι, η εισαγωγή ε, μιας νομικής μορφής για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα επέφερε μια σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό της λειτουργίας των κομμάτων οι κάποιες ε, χώρες ε, δεν θα χρειάζονταν να κάνουν πολλά πράγματα γιατί σε εθνικό επίπεδο ε, πάρα πολλά κόμματα έχουν σαφώς διαμορφωμένη κομματική θέση. Καλό είναι όμως να υπάρξει ε, μία νομική μορφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα κόμματα, η οποία θα πρέπει να είναι απλή και να περιορίζεται σε κάποια τυπικά κριτήρια. Τι είναι το προαπαιτούμενο για να υπάρξει αυτή η νομική θέση. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε και τις εσωτερικές επιπτώσεις μιας τέτοιας διαμόρφωσης ε, νομικής μορφής του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Ε, γιατί ε, και σε εθνικό επίπεδο ε, υπάρχουν ε, διαμορφωμένα κόμματα. Ένα κόμμα βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου τουλάχιστον για τις ευρωεκλογές θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα όπως τα εθνικά πολιτικά κόμματα. Και εδώ υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν και δεν είναι εύκολο πάντα. Εδώ ίσως πρέπει να έχουμε μια ρήτρα μάλλον ευνοουμένου, δηλαδή ότι τουλάχιστον για τις ευρωεκλογέ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται δυσμενέστερα τα ευρωπαϊκά κόμματα από τα εθνικά. Τώρα για τις επιμέρους δραστηριότητες εδώ πρέπει να δούμε κάποια δύσκολα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Δεν είμαι έτοιμος να δώσω ε, περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, ο προσδιορισμός ε, της έννοιας του κόμματος ε, εδώ νομίζω ότι θα με ότι η πολιτική η πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αντικείμενο των συζητήσεων. Πολλές φορές έχουμε ε, ομοσπονδιακές ενώσεις. Τώρα, για τις απαιτήσει. Αναφέρεται η νομική προσωπικότητα, το νομικό πρόσωπο. Ε, ως Γερμανός θα ήθελα να τονίσω ότι τα περισσότερα γερμανικά κόμματα με τη στενή νομική έννοια ε, δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Δεν αποτελούν ε, νομικά πρόσωπα. Με βάση τη νομική, το νομικό καθεστώς μέχρι τώρα θα ήταν δύσκολο τα ευρωπαϊκά κόμματα να έχουν την έδρα τους στη Γερμανία δηλαδή. Και εδώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή νομική μορφή σε εμά. Μια δυσκολία και ένα σημαντικό πρόβλημα βλέπω στις, ε, στα περαιτέρω προαπαιτούμενα για αναγνώριση ενός κόμματος ως ευρωπαϊκού, γιατί απαιτείται να υπάρχει εκπροσώπηση σε χι εθνικά κοινοβούλια και αυτό γιατί είναι προβληματικό. Διότι η πρόσβαση στο εθνικό κοινοβούλιο από κράτος μέλος σε κράτος μέλος παρουσιάζει διαφορές. Έχουμε το όριο του 5%, άλλοι έχουν το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή και είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν χώρες όπου είναι πιο εύκολο να εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από ό,τι σε άλλες χώρες. Άρα πρέπει με μεγάλη προσοχή να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα οι νέες ιδρύσεις κομμάτων ε, είναι ε, ε, ένα άλλο ζήτημα. Ένα τέταρτο των κρατών μελών. Αυτό δεν είναι το μόνο προαπαιτούμενο, υπάρχουν και άλλα που δυσχεραίνουν τη σύσταση ενός νέου κόμματος. Ε, νομίζω ότι οι μέχρι τούδε ισχύοντες κανόνες ε, έχουν κάνει ένα λάθος σε ό,τι αφορά την, τον εντοπισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης ενός κόμματος και την αναγνώριση των προϋποθέσεων για, επιδο, ε, για επιχορηγήσεις δημόσιες ή κρατικές ιδεοδός θεωρούμε ότι ένα κόμμα προέρχεται από τους πολίτες. Πρέπει όμως να φροντίσουμε να ε, μην ε, επεκταθεί αυτό υπέρμετρα. Θα πρέπει να ισχύουν κριτήρια. Δεν μπορεί να απλώνουν όλοι το χέρι και να ε, ζητούν επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό. Επίσης, τα προαπαιτούμενα σε σχέση με τους στόχους των κομμάτων, αυτά ε, δεν αποτελούν πρόβλημα. Για τα ιδρύματα των κομμάτων δεν θέλω να πω πολλά. Ε, μέχρι τώρα προϋποτίθεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ε, ενός ε, τέτοιου ιδρύματος θα πρέπει να έχει περιφερειακή εκπροσώπηση. Αν τα πολιτικά ιδρύματα είναι στενά συνδεδεμένα με κάποιο κόμμα, τότε η υποστήριξη θα πρέπει να προέρχεται κυρίως από το κόμμα, άρα είναι νόμιμο και, τα, και, και, και προϋποτίθεται και τα κόμματα να εκπροσωπούν και περιφέρειες του Νότου για παράδειγμα ή παράκτιες περιφέρειες. Τα κόμματα που εκπροσωπούν τέτοιου είδους συμφέροντα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ε, δημιουργήσουν, να συστήσουν και τέτοιου είδους πολιτικά ιδρύματα. Περνώ στο άλλο βασικό πρόβλημα. Υπό ποιε προϋποθέσεις μπορεί να επιχορηγηθεί ένα κόμμα. Εδώ αποδίδω μεγάλη σημασία στην ισότητα των ευκαιριών. Αναφέρθηκε ήδη πολλές φορές εδώ ότι η πολιτική είναι, ε, σημαίνει ανταγωνισμό. Και ο ανταγωνισμός δεν ε, στηρίζεται μόνο στον ανταγωνισμό ε, συγκεκριμένων μεταξύ συγκεκριμένων ανταγωνιστών, αλλά γίνεται πιο έντονος και πιο αποτελεσματικός, αν λάβει υπόψη δυνητικούς ή δυνάμει ανταγωνιστές. Άρα σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση σε μια αγορά, αν θέλετε. Και σήμερα έχουμε ε, πολλά εμπόδια. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ συγκεκριμένα ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα θέσουμε. Εγώ λέω ότι θα πρέπει τα κριτήρια αυτά να ε, αμβλυνθούν λίγο και τα εμπόδια να χαμηλώσουν. Σημαντικό είναι να έχουμε αυτή την κατανομή των 15%. Τα ε, economies of scale, οικονομίες κλίμακος, ούτως ή άλλως ωφελούν τα μεγάλα κόμματα, οπότε με αυτόν τον κανόνα μπορούμε να έχουμε μια ε, μεγαλύτερη ισότητα των ευκαιριών, είναι καλό αυτό. Επίσης, μέλη, πρόσωπα μέλη των κομμάτων. Βεβαίως, στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ε, τα κόμματα σε αυτό στηρίζονται. Πρέπει όμως να δούμε πολύ ε, προσεκτικά πώς τα ευρωπαϊκά κόμματα μπορεί να εκφράσουν και συνεταιριστικά συμφέροντα. Επίσης, τα κόμματα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά μόνο αν έχουν εσωτερική δημοκρατία. Και αυτό είναι σημαντικό κανόνας. Τώρα, Ποιε νέε μορφές της δημοκρατίας. νέε μορφές δεν χρειάζονται. Οι παλιές καταξιωμένες μορφές είναι ε, αρκετέ. Ε, μυστική ψηφοφορία σε κρίσιμε ψηφοφορίε, εσωτερική δημοκρατία, ε, συνέδρια των αντιπροσώπων, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, επίσης η δημοκρατική διαδικασία στην παρουσίαση και προβολή των ε, υποψηφίων. Ο κύριος Βίλαντ νομίζω ότι ε, έκανε μια σωστή παρέμβαση πάνω σε αυτό το θέμα. Το έκτο ερώτημα αφορά τα, τη σχέση εθνικών προς ευρωπαϊκό κόμματα. Σε ένα πολύ επίπεδο σύστημα όπως το δικό μας, σε περιορισμένο βαθμό έχει νόημα να τραβήξουμε διαχωριστικές γραμμές. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ενοποιητικές γραμμές και αν υπάρχουν συγκρούσεις και εσωκομματικά, ε, η δημοκρατία προσφέρει κανόνες ε, για μια στέρεη αντιπαράθεση ε, και διευθέτηση συγκρούσεων. Δεν είναι κακό να υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών κομματικών μορφωμάτων το ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα ε, μπορούν να χρηματοδοτούνται ε, από το εθνικό επίπεδο, μπορώ να το δεχτώ, ε, πολλά έχουμε δεχτεί από εδώ, αλλά η απαγόρευση έμεσης υποστήριξης για εθνικές προεκλογικές εκστρατείες είναι υπερβολικό. Γιατί να μην είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό κόμμα να μην πει σε εθνική προεκλογική εκστρατεία ότι αυτό είναι αδελφό κόμμα δικό μας, τη δική μας κομματική οικογένεια. Θεωρούμε ότι ε, στην Ευρώπη ασκεί τη σωστή πολιτική ε, και να υποστηριχθεί. Όλα τα άλλα απομακρύνουν από την πολιτική δραστηριότητά τους τα κόμματα και ε, οδηγούν σε λάθος αποτελέσματα. Τώρα για τα δημοψηφίσματα αν με το δημοψήφισμα εννοείται ότι θα γίνει μια ψηφοφορία στα κράτη-μέλη ε, για την συνθήκη, αυτό ε, είναι, υπάρχει δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, ε, βάσει της δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας, έχουμε τώρα το μέσον της πρωτοβουλίας των πολιτών. Η πρωτοβουλία των πολιτών, βέβαια, στηρίζονται σε οργανωτικούς φορείς. Και ποιος είναι ο καλύτερος ενδεδειγμένος ε, τέτοιος φορέας από τα κόμματα. Ε, δεν θέλουμε ε, να παραδοθούμε σε άλλου είδους συμφέροντα, κεφάλαιο κλπ. Γι' αυτό πιστεύω ότι εδώ έχουμε για τα κόμματα έναν τομέα δραστηριοποίησης. Ε, τομέα δραστηριοποίηση των κομμάτων. Αυτό ήταν σημαντικό. Τέτοιου είδου πρωτοβουλίε των πολιτών και οι απορρέουσε από εκεί ε, δραστηριότητε μπορεί να αποτελέσουν ένα τέτοιο τομέα δραστηριότητα. Για το, την ερώτηση 9, ναι, τα κόμματα είναι σημαντική φορείς τη πολιτική διαδικασία και τα πρόσωπα είναι φορείς ταυτότητας ή ταυτοποίησης. Αν θέλω να επιτύχω με τους πολίτες θα πρέπει ε, να ε, βρω πρόσωπα με τα οποία να μπορούν να ταυτίζονται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, ε, προσωπικότητες ε, που θα στέκονται και θα προβάλλονται από τα κόμματα, όπως για παράδειγμα ε, για τους υποψηφίους και το αξίωμα του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η ε, χρηματοδότηση των κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, σωστό, πρέπει να διατηρηθεί, αλλά τα κόμματα μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όταν είναι μέσα και μηχανισμοί που θα μπορούν να αντανακλούν τις δραστηριότητες προς τις ε, εντοπιζόμενες ανάγκες. Ως κόμμα θα ακούσω τον πολίτη όταν μπορώ να πάρω χρήματα και από αυτόν. Εκεί οξύνεται η ακοή. Γι' αυτό μια ίδια χρηματοδότηση σε περιορισμένο βαθμό είναι σωστή. Τέλο για τη χρηματοδότηση μια τελευταία λέξη. Μέχρι τώρα ο κανονισμός δεν γνωρίζει κυρώσει όταν υπάρχουν παραβιάσεις του ε, δημοσιονομικού κανονισμού. Στην πολιτική πολλές φορές όμως ε, παραβιάζονται δικαιώματα, άρα πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται μέχρι τώρα να πρέπει να ανακτώνται τα κονδύλια τα οποία ε, παρατύπωσε δόθησαν. Θα πρέπει να προστίθεται και ένα πρόστιμο εδώ, αλλιώς δεν ωφελεί. Γενικά πιστεύω ότι η ανάπτυξη νομικών προτύπων και κανόνων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας ε, ζωντανής ευρωπαϊκής δημοκρατίας μέσα από τη λειτουργία των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο καθηγητής Μπάρντι, διευθυντής ε, του παρατηρητηρίου για την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Η παρουσίασή μου στηρίζεται σε μια σειρά ερωτήσεων, όπω και του καθηγητή καθηγητού Μόρλοκ, ερωτήσεων που κυκλοφόρησαν σε ένα ερωτηματολόγιο πριν την διεξαγωγή τη ακρόαση. Γι' αυτό και η παρουσίασή μου ουσιαστικά είναι μια σειρά σχολείων παρά μια συγκροτημένη παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για την ε, ίδρυση κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο ζήτημα από νομική άποψη και δεν έχω να προσθέσω και πολλά για τις νομικές πτυχές σε αυτά που ήδη είπε ο καθηγητής Μόρλοκ, γιατί ο καθηγητής Μόρλοκ είναι πλέον η δήμον για τα θέματα αυτά από μένα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να δώσουμε στα ευρωπαϊκά κόμματα και μια νομική προσωπικότητα που θα στηρίζεται στο κοινοτικό δίκαιο. Αν μη τι άλλο, γιατί η νομική αυτή προσωπικότητα θα τους δώσει μεγαλύτερη αίσθηση ταυτότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι που ήδη αναφέρθηκε και το πρωί και συμφωνώ με αυτή την θέση, με αυτή την προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, εμείς και λέω εμείς γιατί ορισμένα από αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και στο παρατηρητηρίο, του οποίου είμαι συνδιευθυντής μαζί με τον Πίτερ Μέγερ. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να απαιτούμε το κόμμα να εκπροσωπείται από, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον από έναν Ευρωβουλευτή. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι τα κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να θεωρούνται ότι συνίστανται από μεμονωμένα στοιχεία συνιστώσεις σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά είναι αλληλένδετες συνιστώσεις ενός ολοκληρωμένου συνόλου. Αν πούμε δηλαδή ότι μόνο κόμματα που έχουν εκλεγμένο ευρωβουλευτή ε, δικαιούνται το χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ουσιαστικά αντιβαίνουμε στην έννοια του κόμματος που κατά τη γνώμη μας είναι σημαντική. Βέβαια αυτό είναι και πολιτικό ζήτημα. Γιατί νομίζουμε ότι έτσι ίσως με, την, ε, το κριτήριο αυτό δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα και ευνοήσουμε περισσότερο τα ήδη γνωστά και καθημερινά ε, κόμματα σε σχέση με τα αναδυόμενα κόμματα, τα νεότερα κόμματα. Αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα και μια πολιτική επιλογή. Δεδομένης της ε, έννοιας και του ορισμού που έχουμε για το Ευρωπαϊκό Κόμμα, πιστεύουμε ότι με μονομένα άτομα, ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γίνουν αν όχι μέλη, τουλάχιστον οπαδοί, υποστηρικτέ και με επίσημο τρόπο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Και εδώ η διάκριση μεταξύ μελών και υποστηρικτών ίσως είναι κάπως λεπτή. Πάντως ε, αυτό που εννοούμε εμείς ότι είναι ότι αυτοί οι υποστηρικτές ή τα μέλη, μονομένα μέλη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, όπως και να τους αποκαλέσουμε τέλος πάντων, δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν ανταγωνισμό με την ιδιότητα μέλους των εθνικών κομμάτων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ιδιότητων. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί λοιπόν ως προς τους δύο αυτούς τρόπους συμμετοχής και να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ό,τι αφορά το θέμα της εσωκομματικής δημοκρατίας και της εσωκομματικής οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι ιδιώτε, τα φυσικά πρόσωπα, οι μεμονωμένοι άνθρωποι που θα γίνουν επίσημα μέλη του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματο, των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων, θα πρέπει να εκλειθούν περισσότερο ω πρέσβει σε εθνικό επίπεδο και υποστηρικτέ περισσότερο, παρά ως ακτιβιστές με την παραδοσιακή έννοια. Βέβαια κάτι τέτοιο και έρχομαι εδώ σε ένα άλλο θέμα, την πέμπτη ερώτηση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να φανεί στην εισαγωγή διαφόρων, διαφόρων μορφών εσωτερικής δημοκρατίας. Αναφέρθηκαν τα συνέδρια, τα κομματικά συνέδρια το πρωί. Αλλά δεν θα τολμούσαμε να συστήσουμε ότι τα συνέδρια κατά το πρότυπο των εθνικών κομματικών συνεδρίων έχουν τέτοιο σκοπό, γιατί τα συνέδρια χάνουν και σημασία και αρχίζουν και υποτιμούνται και σε εθνικό επίπεδο. Θα είμαστε μάλλον υπέρ της αγωγής νέων μορφών εσωτερικής διαβούλευσης, δίνοντας φυσικά συγκεκριμένο βάρος στις διάφορες συνιστώσεις και ακόμη και πριν τις εκλογές. Αυτό είναι πιο δόκιμο κατά τη γνώμη μας, δεδομένη της ε, διάρθρωσης των ε, ευρωπαϊκών κομμάτων. Μία επίσημη ιεραρχική δομή που επιβάλλει ε, μάλλον ε, θεωρεί υπέρτερα τα ευρωπαϊκά κομματικά συνέδρια ως προς τα εθνικά δεν είναι ιδανική κατά τη γνώμη μας μορφή οργανωτική. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο μαζί με τα εθνικά αδελφά κόμματα τους και στις εθνικές προεκλογικές εκστρατείες. Πιστεύουμε δηλαδή ότι κάτι τέτοιο θα ήταν κίνητρο, θα έδινε ενάυσματα για να δημιουργηθεί ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων μορφών πολυεπίπεδης διασύνδεσης που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητη για να δημιουργήσει νέα κόμματα συνεκτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιμένουμε δεν θα πρέπει να θεωρούνται κάτι χωριστό από τα κόμματα σε άλλο επίπεδο. Δύσκολα δηλαδή θα κάναμε διάκριση εμείς μεταξύ των τοπικών ε, και εθνικών κομμάτων εντός του εθνικού κομματικού συστήματος. Και ο λόγος που αναφέρθηκε το πρωί από τη Μόνικα Φρασόνη, ότι αυτός θα ήταν ίσως ο μοναδικός τρόπος για την συμπερίληψη και ευρωπαϊκών ζητημάτων σε εθνικές εκστρατείε είναι πολύ σημαντικό και εύστοχο σχόλιο. Μία άλλη ερώτηση αφορούσε την δυνατότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να χρησιμοποιήσουν κάποιες επιδοτήσεις ή ε, κονδύλια σε εθνικό επίπεδο, στις εθνικές δηλαδή προεκλογικές εκστρατείες. Αυτό θα μπορούσε να προβλεφθεί αρκεί να οριοθετείται σαφώς, ιδιαίτερα προς το ποσοστό των χρησιμοποιούμενων κοινοτικών κονδυλίων για εθνική ό,τι αφορά την ερώτηση των ε, διακρατικών ε, εκλογικών ληστών ή διεθνικών τέτοιων εκλογικών ληστών, πιστεύουμε ότι η ιδέα της θέσπισης μιας διακρατικής ή διεθνικής εκλογικής περιφέρειας είναι μια πιθανή εξέλιξη, μακροπρόθεσμα, αλλά πιστεύουμε ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων και στην οργάνωση των εκστρατιών. Για πρώτη φορά σήμερα το πρωί άκουσα από τον Άντριου Νταφ την πρόταση τη σύσταση, τη ίδρυση μια ειδική κανονιστική υπηρεσία, ενό ειδικού κανονιστικού οργανισμού, ρυθμιστικού οργανισμού. Από πολιτική άποψη ήταν δύσκολο ίσω να προταθεί κάτι τέτοιο και να ιδρυθεί ένα τέτοιο οργανισμό, αλλά νομίζω ότι έχει επίγνωση αυτή τη πολιτική δυσκολία ο κύριο Νταφ. Αλλά η ιδέα δεν μου φαίνεται καθόλου κακή. Σε ό,τι αφορά τι λογικέ συνέπειε της ενίσχυσης του ρόλου των ευρωπαϊκών κομμάτων στις εκστρατείες και στην επιλογή των υποψηφίων σίγουρα θα αυξήσει, ε, θα ενισχύσει το ρόλο τους ό,τι αφορά την δυνατότητά τους να ορίζουν υποψήφιο και για την θέση Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς πιστεύουμε ότι κάθε κόμμα θα πρέπει να προτείνει έναν υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά δεν μπορούμε να προτείνουμε κάτι πιο φιλόδοξο εξαιτία των συνταγματικών όριων. εδώ η δημιουργία ενός πολιτικού ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με την αύξηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην εκτελεστική εξουσία, στα εκτελεστικά όργανα. Κάτι τέτοιο φυσικά θα απαιτούσε προηγούμενη μεταρρύθμιση που είναι μάλλον απίθανο να λάβει χώρα στο εγγύς μέλλον. Εν κατακλείδη θα μπορούσα να πω ότι το κριτήριο της αυτοχρηματοδότησης θα μπορούσε να διατηρηθεί, μια και είναι ένα στοιχείο για την ολοκλήρωση των κομμάτων σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η προσέγγιση που αντιμετωπίζει τα ως ξεχωριστές οντότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι ασύμβατη με οποιαδήποτε έννοια κόμματο που έχουμε και σε ομοσπονδιακό αλλά και σε μη ομοσπονδιακό εθνικό σύστημα. Δεν νοείται τέτοια διάκριση, τέτοιος διαχωρισμός όπως μερικές φορές ακούμε να απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς αυτό τονίζεται και από το διτό χαρακτήρα, τον υπερεθνικό και τον διακρατικό της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, της διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε μόνο με μια αναθεώρηση του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ενίσχυε την υπερεθνική της διάσταση. Γνωρίζουμε όμως ότι και τέτοιου είδους αναθεώρηση και τέτοιου είδους προοπτική είναι μάλλον απίθανη για το εγγύς μέλλον. Βέβαια, χωρίς κάτι τέτοιο, τα, το σύστημα ευρωπαϊκών κομμάτων έχει κάποια όρια. Και εκεί είναι πολύ, θα τα συναντήσει πολύ σύντομα αυτά τα όρια. Όσο και αν βελτιώσουμε το σύστημα ευρωπαϊκών κομμάτων, ε, πιστεύουμε ότι είναι αδιανόητο ένα κβαντικό άλμα στις εξελίξεις του και στην δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος ευρωπαϊκών κομμάτων. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να είναι συγκροτημένο αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πολιτικών Κομμάτων, προκειμένου να προωθεί την ολοκλήρωση των κομματικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα και διαφυλάσσοντας την αυτονομία σε όλα τα επίπεδα και στα μεμονωμένα κόμματα, αλλά και δίνοντας ενάυσματα για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των συνιστοσών σε όλα τα επίπεδα, μπορούμε μόνο με αυτόν τον τρόπο να ελπίζουμε σε ένα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 να εκφράσω καταρχήν τις θερμές μου ευχαριστίες ε, στην Συνταγματική Επιτροπή που με κάλεσε να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση και ειδικότερα προς την εισηγήτρια της Επιτροπής, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία συνέταξε μία έκθεση η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης αλλά και μία πρόκληση για μία ζωηρή συζήτηση για την εξέλιξη των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη μια συζήτηση η οποία λαμβάνει χώρα ε, σε έναν χώρο που θεωρείται την πιο, ως η πιο σύνθετη πολιτεία που έχει ποτέ συσταθεί. Τώρα, αν αυτή είναι μια συμπολιτεία, για να αναφερθώ στον ε, καθηγητή Τσάτσον, ή αν είναι μια ε, συγκυριαρχία, Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προβολή ε, μιας, ε, ε, ενός συνδυασμού δημοκρατικών πολιτιών ή πολιτικών μορφωμάτων σε ό,τι αφορά την κοινή άσκηση των εξουσιών και νομίζω ότι έτσι κινούμεθα προς μια σύνθετη δημοκρατική τάξη. Όμως ο σχεδιασμός ενός μεταρρυθμιστικού πακέτου για τα ευρωπαϊκά κόμματα ως μέσον κινητοποίησης δημοκρατικών δυναμικών των μεμονωμένων και οργανωμένων πολιτών δεν είναι εύκολη υπόθεση και σίγουρα προϋποθέτει ε, μια διευκρίνηση της αποστολής των ευρωπαϊκών κομμάτων από την ε, ίδρυσή τους και μετά και πώς μπορεί να λάβει χώρα ένας ενημερωμένος ε, διάλογος βάσει αρχών για να δημιουργήσει και να οδηγήσει στην ανάδυση ενός Δήμου στον πληθυντικό των Δήμων. Υπάρχουν πολλές ασυμμετρίες, ε, υπάρχει το πρόβλημα της αυξανόμενης ε, ε, αποχής, το αποθαρρυντικό επίπεδο της ταύτισης των πολιτών με τα κόμματα. Τα ευρωπαϊκά κόμματα είναι πολύ σημαντικά για την βελτίωση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Όχι μόνο ε, με βάση αυτό που έγραψε ο Σατ Σνάιντερ πριν από 60-70 χρόνια, που είπε ότι τα πολιτικά κόμματα δημιούργησαν τη σύγχρονη δημοκρατία και η σύγχρονη δημοκρατία είναι αδιανόητη, εκτός και αν λειτουργεί μέσα από τα πολιτικά κόμματα, αλλά και, ε, όπως αναφέρεται και από την κυρία Γιαννάκου, τα πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα συμβάλλουν στην διαμόρφωση θέλησης, ε, διότι συμβάλλουν ε, στην ε, θέσμιση της ε, κοινωνίας. Τα ευρωπαϊκά κόμματα μπορεί να λειτουργούν ως παράγοντες συστημικής αλλαγής, διευκολύνοντας την δημιουργία νέων πολιτικών ταυτοποιήσεων, μπορούν να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν την ε, πολιτικοποίηση να δημιουργήσουν ένα κομματικό σύστημα ε, καινούριο και πάνω απ' όλα να δώσουν στους Ευρωπαίους πολίτες μια αίσθηση του ανήκειν σε Δήμο. Ε, έτσι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει μια δημοκρατική πορεία γενικότερα με βάση τον Δήμο με την αρχαία ελληνική έννοια. Πώς θα συγκροτηθεί και θα διατηρηθεί ένας Δήμος Μπορεί τα ευρωπαϊκά κόμματα να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας ε, ταυτότητας του πολίτη και να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας πολιτικής ευρωπαϊκής συνείδησης και να εκφράσουν την πολιτική βούληση των πολιτών της Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κόμματα να επικεντρωθούν πλέον τώρα όχι μόνο σε ερωτήματα του ποιος κυβερνά και πώς, αλλά, αυτό μπορεί να είναι πιο σημαντικό, ποιος κυβερνάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προϋποθέτει μία δομημένη συζήτηση, αντιπαράθεση, σχετικά με το ποιο Δήμο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, τα οποία ε, με βάση τον Πέτιτς ε, ε, θα πρέπει να ακολουθούν ε, τρόπους διαβουλεύεσθε και τη μέθοδο του διαβουλεύεσθε για την λήψη των αποφάσεων περιλαμβάνοντας όλες τις σημαντικές φωνές διαφοράς μέσα στην κοινότητα. Έτσι θα πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει ελευθερία ανάπτυξης κοινών δημοκρατικών βάσεων για να επιδιωχθούν πολιτικοί στόχοι. Έτσι λοιπόν πολλοί λαοί ένας δήμος παρά ε, δίνει ένας λαός αυτό ε, νομίζω ότι προσελκύει την φαντασία ε, και θα μπορούσαμε έτσι να φτάσουμε σε ένα δήμο στον πληθυντικό. Ε, η νομική θέση και η νομική προσωπικότητα θα μπορούσε να μην στηρίζεται τόσο πολύ στους στα εθνικά αντίστοιχα κόμματα, ε, ε, αντίθετα θα μπορούσαν να δράσουν ως αντιπροσωπευτικοί φορείς των, ευρωπαϊκών πολιτικών συμφερόντων τα ευρωπαϊκά κόμματα. Αυτό ε, θα επέτρεπε να δημιουργηθεί ένα και θα βελτίωνε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά κόμματα, θα μπορούσαν έτσι να έχουν και μια πλατφόρμα για να μπορέσουν να ενισχύσουν και να σφυριλατήσουν ακόμα πιο στενούς εκλογικούς και καθημερινούς δεσμούς με τους πολίτες. Τα ευρωπαϊκά κόμματα θα μπορούσαν έτσι να εισαγάγουν καινοτόμα μέσα για να συνδέονται με την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη μια διεθνική ε, κομματική λίστα θα ήταν καλό διότι θα μπορούσαν να προβάλλονται υποψήφοι οι οποίοι εκπροσωπούν γνήσια ευρωπαϊκά θέματα και πολιτικές πλατφόρμες αντί να ανταγωνίζονται για την ε, ψήφο του λαού σε προεκλογικές εκστρατείες αποσπασματικές, χαμηλού προφίλ, υποτιμημένες, υποδέστερες ε, που αντικατοπτρίζουν μόνο εθνικά, εθνικές ατζέντες. Ε, επίσης το θέμα των ε, ε, δημοψηφισμάτων είναι ένα θέμα το οποίο οδηγεί σε μια σειρά από προκλήσεις για την πολιτική, συλλογική πολιτική ικανότητά τους να αρθρώσουν πολιτικό λόγο μέσα προς τους πολίτες. Ε, αυτά τα δημοψηφίσματα θα συνδέονταν άμεσα προς ε, την ενωσιακή πολιτική, αλλά επειδή ως διαμορφωτές της πολιτικής βούλησης τα ευρωπαϊκά κόμματα δικαιούνται να λειτουργούν ως πολιτικοί εκπαιδευτές ε, που μπορούν να καθορίζουν την συμβίωση των πολιτών μέσα σε μια ευρύτερη πολιτεία ρύθμιση των ευρωπαϊκών κομμάτων είναι ένα ε, μέρος ευρύτερης εξέλιξης του, της νομοθεσίας για τα πολιτικά κόμματα. Ο Σάιμον Χίξε λέει ότι η ε, ευρωπαϊκή πολιτεία είναι μια πολιτεία όπως οποιαδήποτε άλλη και η οποία λαμβάνει υπόψη διάφορες αντιλήψεις για την ευρωδημοκρατία που μπορεί να είναι από μια μεταεθνική απόψη σχετικά με το κράτος του Δήμου ή το, το κράτος ενός Δήμου, Δημοσκρασί ή προς πιο ε, μηχανιστικές, κράτοκεντρικές αντιλήψεις ε, για το κράτος πολλών Δήμων. Από την προηγούμενη άποψη που είναι το θεσμοθετημένο ισοδύναμο ε, διαφορετικών πολιτών που διαμορφώνουν το μέλλον τους από κοινού, μπορεί ε, το καταστατικό ενός Ευρωπαϊκού Κόμματος να οδηγήσει σε μια νομική θέση και προσωπικότητα ευρωκομμάτων που ε, μπορούν να δράσουν ως παράγοντες της, πολιτικής, της διαμόρφωσης πολιτικής βούλησης σε επίπεδο ένωσης. Από την άλλη πλευρά, το κράτος πολλών δήμων προβλέπει ένα μινιμαλιστικό ή λειτουργικό ρόλο, πιο περιοριστικό για τα κόμματα, για τα, τα ευρωπαϊκά κόμματα, ε, ως μια προέκταση των ε, εθνικών κομματικών δομών και μορφών πολιτικής ε, προβολής ή αντιπαράθεσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να χειριστούμε τα πολλαπλά και πολλαπλασιαζόμενα δημοκρατικά ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καταστατικό ενός Ευρωπαϊκού Κόμματος ε, έχει ρόλο να παίξει αντιμετωπίζοντας τα χαμηλά επίπεδα ε, διαμόρφωσης ε, της συνείδησης του πολίτη μεταξύ των Ευρωπαίων. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για μια τέτοια μεταρρύθμιση. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ και οι πιο εκλεπτισμένες ε, και οι λεπτομέρειες της ε, παρέμβασής μου υπάρχουν γραπτός, ε, μπορούν να οδηγήσουν σε αντιμετώπιση της ετερογένειας από τους πολίτες που τώρα είναι μια συνθήκη για την Ένωση, όχι ενοποίηση ε, ευρύτερων ε, ομάδων ευρωπαϊκών πληθυσμών που έχουν, ε, αν θέλετε, την αντίληψη Caritas Republicae, η αγάπη για όλα τα κοινά ή τα ευρωπαϊκά θέματα μέσα σε μια ευρύτερη πολιτεία, που με βάση τον Ιγνάτιεφ ε, φιλόδοξη να γίνει μια κοινότητα ενωμένη σε ένα κοινό επιχείρημα σχετικά με το νόημα, το εύρος ε, της ελευθερίας. Η Ευρώπη όμως για να μπορεί να, αποτελέσει έναν Δήμο θα πρέπει να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά κόμματα ε, οικοδομώντας πάνω σε διεθνικά δικαιώματα και ε, διαμορφώνοντας το κατάλληλο κομματικό σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι θα πρέπει να αντιδρά καλύτερα στο εκλογικό σώμα και τις ανάγκες του για να ε, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ε, Δήμου με των πολιτών. Είναι σημαντικό να ε, ε, να υπάρξει μια κατανομή ε, δικαιωμάτων και αρχών και αξιών στην αναδιόμενη αυτή κοινωνία των πολιτών προσφέροντας μια αίσθηση προσανατολισμού που θα μπορέσει να εμπνεύσει τους πολίτες υπέρ του Δήμου. Ευχαριστώ καθηγητά. Πραγματικά είμαστε στην ώρα μας και μπορούμε με ηρεμία να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Πριν ε, ολοκληρώνουμε μετά στη συνέχεια με τις ε, τοποθετήσεις του δόκτωρα Γκάλερ ανάλυση για τη χρηματοδότηση και την οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων και τελειώσαμε. Α, και μετά έχουμε και την διαφάνεια. Η κυρία Μίτερ Μάιερ. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση για αυτές τις ε, τρεις πρώτες εισηγήσει. Ζήτησαν το λόγο ο συνάδελφος Χέφνερ και ο συνάδελφος Ρανζέλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις των τριών εμπειρογνωμόνων μας. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Πρέπει να θέσουμε κανόνες. Χρειάζονται περισσότερες αντιπαραθέσει συζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζονται οι παράγοντες για αυτό το πράγμα και γι' αυτό χρειάζονται τα ευρωπαϊκά κόμματα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τωρινή μας απόφαση το τι θα ε, ισχύσει στο μέλλον. Υπάρχει ένας κίνδυνος, πάντα υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος να νομοθετεί κανείς ε, κοιτάζοντας περισσότερο ίδια ε, ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν τις ρυθμίσεις να μην τις επιλέξουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία εξουσία μας, αλλά να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ε, δημοκρατική εμφισβήτηση των εξουσιών που θα θεσπίσουμε. Παλαιότερα τα παιδιά ε, είχαν μεγαλύτερη ελευθερία να παίζουν και σκαρφάλωναν σε λόφους ε, θέλοντας να κατακτήσουν την κορυφή. Αν πούμε τώρα ότι ε, το, το, στο Ευρωπαϊκό Κόμμα θα μπορεί να μετέχει μόνο όποιο είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό δεν είναι πολύ ευρωπαϊκή ιδέα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ερωτηθούν εκείνοι που τάσσονται υπέρ αυτή τη προσέγγισης πώς θα αντιμετωπίσουν την πολιτική αλλαγή. Όχι μόνο στους κόλπους των κομμάτων, αλλά αλλαγή με την έννοια νέε ιδέε, νέα κόμματα που θα διαμορφωθούν, θα αποκρισταλωθούν και θα οδηγήσουν ε, σε αλλαγή του κομματικού τοπίου. Αυτό δυνάμει είναι ε, πιθανό. Χρειάζεται λοιπόν μια νομική μορφή η οποία δεν θα εξυπηρετεί κάτι άλλο ώστε να είναι ακατάλληλη ε, η βέλγικη μορφή non-profit μη κερδοσκοπική οργάνωση, αλλά θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη νομική μορφή, χωρίς να την περιορίζουμε σε αυτούς που σήμερα είναι ισχυροί. Θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία, πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση σε ανθρώπους που θα θελήσουν να δημιουργήσουν, να ιδρύσουν ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Θα πρέπει να δούμε όμως αν ένα τέτοιο συνασπισμό πολιτών πληρεί τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να χρηματοδοτείται, να χρηματοδοτείται η προεκλογική εκστρατεία του να χρηματοδοτείται η λειτουργία, η τήρηση, η διατήρηση γραφείων κλπ. Όλα αυτά συνδέονται με άλλες προϋποθέσεις. Ότι δηλαδή θα πρέπει κανείς να έχει σημειώσει κάποια πρόοδο, κάποια επιτυχία και να μπορεί έτσι να αποδείξει ότι υπάρχει ένας ικανός αριθμός πολιτών που στηρίζουν αυτή την πολιτική δύναμη και ότι στην προεκλογική εκστρατεία παρουσιάζεται και προβάλλει αρκετό ικανό αριθμό υποψηφίων ε, προτάσεων προγραμμάτων. Τώρα, πώς θα μπορούσαμε να βοηθηθούμε, μπορούμε να, τα, να κάνουμε διαχωρισμούς. Εδώ είναι κάτι σημαντικό που μπορεί να προκύψει ο συμπέρασμα αυτή τη ακρόαση, Ότι δηλαδή δεν είναι σωστό η νομική μορφή του πολιτικού κόμματος και η χρηματοδότηση του πολιτικού κόμματος να είναι ασύνδετες. Αν αποσυνδεθούν, καλό θα ήταν να υποβάλλουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, τι νομικές και ε, ε, άλλες προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύσουν. Επίσης, ε, πολλοί ανέφεραν και ο συνάδελφος Βίλαντ στο τέλος. Είπαν ότι εμείς θα πρέπει να αξιώσουμε το Ευρωπαϊκό Κόμμα το οποίο συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και στις ευρωπαϊκές εκλογές να είναι το ίδιο δημοκρατικό. Άρα, αν υπάρχουν κόμματα τα οποία ορίζουν τους ε, υποψηφίους με τρόπο αντιδημοκρατικό ή μυστικό, Αυτά τα κόμματα δεν πρέπει να αναγνωρίζονται. Ε, αυτά είναι τα βασικά σημεία που ήθελα να θέσω. Επίσης, ένα άλλο δύσκολο θέμα είναι η σχέση με μεμονωμένων μελών και εθνικών ή περιφερειακών κομμάτων. Πιστεύω ότι χρειάζονται και τα δύο. Ε, στους για παράδειγμα. Ε, υπάρχουν ε, κόμματα που δημιουργήθηκαν από ε, συνασπισμούς σε εθνικό επίπεδο. Και μπορεί κάποιος να πει, εγώ θέλω να προσχωρήσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εργαστώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα. Αυτό όμως ανοίγει πολλά προβλήματα σε σχέση με την ισορροπία μεταξύ τους. Σήμερα το πρωί άκουσα πολλές παρεμβάσεις που τάχθηκαν υπέρ της μιας ή της άλλης λύσης θα ήμουν ευγνώμων να συζητήσω, αν μπορούσαμε να συζητήσουμε περισσότερο για τη νομική ε, πλευρά του θέματος και πώς μπορούμε με επιτυχή τρόπο και λειτουργικό τρόπο να συγκεράσουμε τα δύο επίπεδα. Περιορίζομαι σε αυτές τις ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι εδώ έχουμε μια ευκαιρία να συμβάλλουμε πολύ σημαντικά ε, στην ευρωπαϊκή δημοκρατία αν μεταξύ άλλων αντισταθούμε στον πειρασμό να περιοριστούμε στα ίδια συμφέροντα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο την ποικιλομορφία στην Ευρώπη, ούτω ώστε να λειτουργεί όσο γίνεται καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ραζέλ. Θα ήθελα να υποβάλω τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις ή μάλλον σχόλια καλύτερα και να υποβάλω και μια-δυο ερωτήσεις. Πιστεύω καταρχήν, όπως είπε ο κύριος Χέφνερ, θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το νομικό ή κανονιστικό καθεστώς των πολιτικών κομμάτων και να επιλύσουμε και το ζήτημα της χρηματοδότησης. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δεχθούμε την ύπαρξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τη χρηματοδότηση να την κρατήσουμε μόνο για ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που θα έχουν εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, παρόμοιο σύστημα ισχύει σε ορισμένες χώρες. Και νομίζω ότι είναι αρκετά ισορροπημένο. γιατί επιτρέπουμε την πρόσβαση των πολιτών και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κόμματος, αλλά θεσπίζουμε το εχέγγυο ότι μπορούν να αξιοποιήσουν την κοινοτική χρηματοδότηση μόνο εφόσον αποδείξουν ότι έχουν κάποια ευρωπαϊκή σημασία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κριτήριο για να διαθετήσουμε το ζήτημα της χρηματοδότησης. Μία άλλη παρατήρηση που είναι σημαντική αφορά το θέμα της, του μέλους, της ιδιότητας του μέλους. Αυτό είναι όντως περίπλοκο θέμα, αλλά θα πρέπει να δεχτούμε, πιστεύω ρητά, ότι με μεμονωμένη ε, ιδιότητα μέλους είναι πολύ σημαντική. Ατομική ιδιότητα μέλους. Υπάρχουν άλλωστε προηγούμενα περιπτώσεις που ίσως δεν αναφέρονται εδώ, αλλά εγώ θυμάμαι την περίπτωση ενός ευρωβουλευτή, του Λούκα Πύρες, πολύ γνωστού εδώ, Πορτογάλου ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ήταν μέλος του CDS, που τώρα είναι ε, πολιτικό κόμμα, αριστερό, αλλά και προευρωπαϊκό. Ε, επειδή ήταν πολύ φιλοευρωπαϊστής ο κύριος Λούκας Πύρες, άφησε το κόμμα του στην Πορτογαλία και έγινε μέλος του ΕΛΚ. Εξελέγει ε, στο PSD, που είναι μέλος του ΕΛΚ, και έτσι για ένα διάστημα ήταν μέλος του ΕΛΚ, αλλά δεν ήταν μέλος του PSD, γιατί άφησε το PSD. Οπότε θα υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα και άλλων που μπορεί να είναι ανθρώπων που είναι μέλη ενός Ευρωπαϊκού Κόμματος, αλλά δεν θέλουν ταυτόχρονα να θεωρούνται και μέλη του δι... εθνικού τους κόμματος. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Είχαμε μία περίπτωση αυτή που σας ανέφερα του κυρίου Λουκασπύρες, αλλά μας δείχνει μία τέτοια περίπτωση ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμε και την ατομική ιδιότητα μέλους. Ένα Μία πιθανή λύση θα ήταν να πούμε ότι όλα τα μέλη των εθνικών κομμάτων είναι αυτομάτως και μέλη του Ευρωπαϊκού Κόμματος, αλλά υπάρχει και δυνατότητα να είναι κανείς μέλος ενός Ευρωπαϊκού Κόμματος, χωρίς ταυτόχρονα να είναι και μέλος του Εθνικού του Κόμματος, ενός Εθνικού Κόμματος. Αυτή θα ήταν μια μεικτή λύση, μια συνδυασμένη λύση. Και φυσικά διαφυλάσσουμε και το συνταγματικό ε, δικαίωμα να είναι κανείς μέλος ενός εθνικού κόμματος χωρίς να είναι και μέλος ενός ευρωπαϊκού κόμματος κατά ανάγκη. Αλλά να το πούμε ρητά, να προβλέψουμε και αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ευρωπαϊκή ιδέα, για το ευρωπαϊκό ιδεώδες και για το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε αυτή την συνείδηση της ατομικής ιδιότητας μέλους. Και υπάρχει νομίζω δυνατότητα, υπάρχει περιθώριο για πολλούς που πολύ πιθανό να θέλουν να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αλλά έχουν δυσκολίες ή είναι απρόθυμοι να ανήκουν και σε εθνικά κόμματα. Η τρίτη μου παρατήρηση αφορά άμεσα ένα θέμα που είχαμε συζητήσει πριν ακούσουμε τις απογευματινές ομιλίες, το θέμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δυνατότητα υποβολής υποψηφίου ε, που μπορεί να κατεβαίνει ως ε, υποψήφιος ενός κόμματος στις ευρωεκλογέ. Αυτό είναι αρκετά περίπλοκο ζήτημα. Γιατί Κάτι τέτοιο θα άλλαζε το πολιτικό σύστημα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και έρχομαι στις ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι υποψήφιος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται στο Βρετανικό σύστημα. Αν θέλει κανείς να είναι πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι και μέλος του Κοινοβουλίου. Ακόμη και αν μετά παρετηθεί από την ιδιότητα του βουλευτή και μεταβεί στην Επιτροπή. Ερώτηση κάνω. Αν έχουμε έναν υποψήφιο που δεν είναι υποψήφιος του Κοινοβουλίου, μπορεί να είναι μόνο υποψήφιος ε, της Ευρωπα... για τη θέση Πρόεδρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι και υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να εκλέγουμε άμεσα τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα είναι το πολιτικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας πρότασης, τότε θα διαμορφώσουμε ένα είδος προεδρικού συστήματος και όχι κοινοβουλευτικού. Επίσης, έχουμε και, μια πολύ δύσκολη σχέση, ένα πολύ, μια πολύ δύσκολη σχέση μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου. Γιατί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν έχει άμεση δημοκρατική νομοποίηση θα ανταγωνίζεται ουσιαστικά τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Και μάλιστα με πολύ σκληρό τρόπο. Δεν λέω ότι κατά ανάγκη αυτό είναι κακό. Αλλά λέω ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα συμβεί αν δεχτούμε μια τέτοια πρόταση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το είδος του πολιτικού συστήματος που επιθυμούμε. Και αν αλλάξουμε μόνο το εκλογικό σύστημα ή το κομματικό σύστημα, δεν πρόκειται να αλλάξουμε όλο το σύστημα ελέγχων και παληθεύσεων του συνολικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος. Αυτό βέβαια δεν είναι τραγικό, το αντίθετο. Εγώ Είμαι υπέρμαχος της συνταγματικής εξέλιξης και μπορούμε να επιφέρουμε συνταγματικές αναθεωρήσεις χωρίς να τις χαρακτηρίζουμε και τέτοιες. Αλλά αυτό θα συμβεί αν ξεκινήσουμε μια διαδικασία όπου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εκλέγεται άμεσα. Είτε είναι μέλος του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε όχι. Αν εκλέγεται άμεσα, τότε θα δημιουργηθούν ε, παραλληλισμοί με το αμερικανικό σύστημα. Έχουμε και τον πρόεδρο της Γερουσίας, που είναι ο πρόεδρος του, πρόεδρο του Συμβουλίου δηλαδή, που θα βρεθεί σε πολύ περίεργη θέση. Αλλά είναι πολύ θα, βρεθεί σε ένα πολύ δημιουργικό και καινοτόμο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, να εξετάσουμε τις συνέπειες ενός, ε, μιας κομματικής λίστας που θα περιλαμβάνει και ένα συγκεκριμένο υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό ήταν κάπως παράδοξο, περίεργο, γιατί τότε θα είχαμε τη δυνατότητα να εκλέγει ο Ευρωπαίος πολίτης τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα είχαμε ταυτόχρονα και ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μπορεί να υποχρεώσει σε παρέτηση τον πρόεδρο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς είναι δυνατόν ε, ένα κοινοβούλιο να εκφράσει μορφή έλλειψη εμπιστοσύνη ή δυσπιστία σε ένα πρόεδρο που έχει εκλεγεί άμεσα όμω από του Ευρωπαίου πολίτε. Νοείται κάτι τέτοιο. Είναι δυνατό σε περίπτωση διάπραξη ενό εγκλήματο, για παράδειγμα. Στι Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αλλά είναι απαράδεκτο ο πρόεδρο εκτελεστικού σώματος να ε, ε, εξαναγκάζεται σε, παράτα, σε παρέτηση από ένα κοινοβουλευτικό σώμα ενώ έχει εκλεγεί άμεσα με τη λαϊκή τιμιγορία. Αυτό είναι κάπως περίεργο. Αυτή η κατάσταση που θα δημιουργηθεί θα είναι κάπως περίεργη. Γι' αυτό θα πρέπει να προβληματιστούμε περισσότερο και να αναλύσουμε πιο διεξοδικά όλες τις συνέπειες μιας τέτοιας πρότασης. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αρκετά σας προβλημάτισα. Νομίζω ότι αρκετή τροφή για συζήτηση έδωσα. Ευχαριστώ. Ε, Είχα ζητήσει αρχικά το λόγο για κάτι όμως ε, που ανέφεραν οι συνάδελφοι και με κάλυψαν. Είναι σκόπιμο να γίνει μια διάκριση μεταξύ της ρύθμισης της ύπαρξης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από την δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Και όταν λέω να γίνει διάκριση, διαχωρισμός, εννοώ να προβλεφθούν διαφορετικές προϋποθέσεις. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει καμία σύνδεση, αλλά έχει νόημα, είναι σκόπιμο για τη δημιουργία ενός νομικού καθεστώτος που θα αναγνωρίζει ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, να απαιτούμε μια σειρά προϋποθέσεων, για παράδειγμα να υπάρχουν εκπρόσωποι πολλών ε, χωρών ή να πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων πολλών χωρών ή τοπικών κομμάτων. Αλλά για τη χρηματοδότηση, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και δεν πρόκειται να επιμείνω και εγώ άλλο σε αυτό, απαιτείται όπως συμβαίνει και στις ε, περιπτώσεις κρατικής χρηματοδότησης πολλών χωρών και στην Ισπανία για παράδειγμα, είναι απαραίτητο για να δικαιούται κανείς τέτοια δημόσια χρηματοδότηση να έχει εκπροσώπηση μετά από εκλογές. Δηλαδή οι πολίτες να έχουν δώσει την υποστήριξή τους, ένα επίπεδο υποστήριξης σε αυτά τα κόμματα και αυτή η υποστήριξη να φαίνεται από την παρουσία τους ε, σε, ε, είτε σε Εθνικό Κοινοβούλιο, είτε σε τοπικά κοινοβούλια και σε περίπτωση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων να φαίνεται η εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη γνώμη μου είναι αδιανόητο να θεσπίσουμε κοινοτική χρηματοδότηση την οποία θα δικαιούται ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που δεν θα έχει κανέναν απολύτω ε, ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα έχει καμία εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντίθετα μπορώ κάλλιστα να φανταστώ την ύπαρξη ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που είναι σε φάση ίδρυσης ε, ή ανάπτυξης, αλλά δεν έχουν ε, κατακτήσει ακόμη ένα επίπεδο εκπροσώπησης που να τις ε, καθιστά επιλέξιμες για κοινωτική χρηματοδότηση. Όπως είπε ο κύριος Ρανζέλ, και είναι, ήταν πολύ εύστοχες και μεστές οι παρατηρήσεις του, αλλά δεν νομίζω ότι επηρεάζουν το θέμα της ρύθμισης του νομικού καθεστώτος των κομμάτων. Τουλάχιστον δεν επηρεάζουν άμεσα αυτό το καθεστώς. Γιατί εδώ προσπαθούμε να ορίσουμε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, να θεσπίσουμε τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν, τους όρους της χρηματοδότησης. Κάποια στιγμή μπορεί να ανακύψει το θέμα του κατά πόσο μία από τις λειτουργίες αυτών των κομμάτων θα είναι να καταρτήσουν και διεθνικούς, υπερεθνικούς ε, καταλόγους ή υπερεθνικές εκλογικές λίστες που θα περιλαμβάνουν και τον υποψήφιο ε, της ε, Ευρωπαϊκής, στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση που θα συγκεντρώσουν την πλειοψηφία στις ευρωεκλογέ. Αλλά στο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα για τη συζήτηση της έκθεσης Γιαννάκου, δεν νομίζω ότι ε, έχει ακόμη οριμάσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν έχει καν τεθεί αυτό το θέμα αυτό. Αυτό έχει τεθεί από πρωτοβουλίες κάποιων κομμάτων. Ε, μεταξύ άλλων και, κομμά... και πρωτοβουλίες των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η σύγκριση που έκανε ο κύριος Ρανζέλ με διάφορες χώρες, οι κράτη-μέλη της Ένωσης, δεν οδηγεί σε λύσεις παρά μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Είμαστε ένα μόρφωμα sui generis, όπως αναφέρεται και από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Υπάρχει κράτος μέλος όπου άμεσα εκλεγμένος πρόεδρος στο άμεσα εκλεγμένο κοινοβούλιο ε, μπορεί ε, να αλληλεπιδράσει και να λειτουργήσει. Ή, ε, υπάρχουν δηλαδή πολύ προηγμένα ε, συστήματα λειτουργίας της δημοκρατίας. Θα πρέπει να δούμε εμείς πώς, τι συνέχεια μπορούμε να δώσουμε. Αυτό που θα έπρεπε είναι ότι στα επόμενά μας βήματα θα πρέπει να περιοριστούμε, να αυτοπεριοριστούμε ε, στα πλαίσια που έχουμε διαμορφώσει. Δηλαδή, να θεωρήσουμε ότι άμεσα δεν θα υπάρξει τροποποίηση της συνθήκης και θα πρέπει να κάνουμε αυτά που μας επιτρέπει η συνθήκη. Ε, το ε, θέμα το, της ημέρας των εκλογών, Πέμπτη, Κυριακή ή τον εκλογικό νόμο. Μέχρι τώρα, μέχρι την αλλαγή του, της κυβέρνησης στη Βρετανία υπήρχαν ε, διαφορές στον εκλογικό νόμο. Υπάρχουν ε, πολλές πρακτικές που αποφεύγονται σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, ενώ όχι σε άλλα. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε τι μέσα διαθέτουμε και τι πλαίσια διαθέτουμε. Θα πρέπει να περιοριστούμε, όπως σας είπα, σε αυτά που δεν προϋποθέτουν ε, τροποποίηση της συνθήκης. Ε, ένα πράγμα που δεν με ικανοποιεί και αναφέρθηκε από τους δύο τελευταίους ομιλητές, τι θα κάνουμε με τους επιτρόπους που θέλουν να είναι υποψήφιοι. Δηλαδή, ε, έξι μήνες πριν από την εκλογή να παρετούνται για να γίνουν υποψήφοι ε, ευρωβουλευτές και μετά να ξαναγίνουν επίτροποι. Δηλαδή αυτό είναι ένα σύστημα δυσχερές, το οποίο δεν θα γίνει κατανοητό από τους πολίτες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αλλαγή όταν θέλουμε να βάλουμε τον επικεφαλής, να ορίσουμε και να προβάλλουμε τον επικεφαλής υποψήφιο. Δηλαδή, μια οικογένεια κομμάτων μπορεί να προβάλλει έναν υποψήφιο, τον κεντρικό υποψήφιο. Αυτό παίζει, ε, ε, αυτό που θα κρίνει είναι η αποδοχή του κόμματος από τους πολίτες. Θα πρέπει δηλαδή να έχω ε, ορισμένες διασφαλίσεις για να το κάνω αυτό. Και από πολιτικής άποψης η δύναμη των κομμάτων μπορεί να καθορίσει και τον υποψήφιο που μπορεί να είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής. Εάν ε, κάποια κόμματα ε, αποφασίσουν να δεχτούν τον ε, κεντρικό τους υποψήφιο, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή τη γνώμη. Όποιος υποψήφιος δεν έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία θα σκεφτεί πολύ προσεκτικά θα σκεφτεί δύο φορές εάν θα περάσει ως επικεφαλής σε εισαγωγικά της αντιπολίτευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, αποφασίζονται με το σωστό τρόπο οι υποψήφοι, δηλαδή να υπάρξουν κάποιοι αυτοματισμοί ε, που θα ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή και τροποποίηση. Επίση, η Κομισιόν ε, ανέφερε πριν από λίγο καιρό και αυτό το ε, ήλεγξε ο Γερμανός ε, Επίτροπος αν δηλαδή μπορεί να είναι και μπορεί να παραμείνει ενεργό μέλος ενός κόμματος ή αν θα πρέπει να απαρατηθεί από την ιδιότητα του μέλους όπως ο Γερμανός Πρόεδρος Νομίζω ότι δεν πρέπει να ευνουχίζουμε πολιτικά τους επιτρόπους στη χώρα καταγωγής τους, ανεξάρτητα από το ποια είναι αυτή. Άρα θα πρέπει να δούμε εάν κάποιος μπορεί να, ε, να δούμε ποια είναι η διαδικασία μέσα από την οποία μπορεί ένας επίτροπος να υποβάλει υποψηφιότητα για ε, την Ευρωβουλή. Δεν πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές. Ε, σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο ισχύει και για το εσωτερικό των κομμάτων, γιατί πράγματι έχουμε και εδώ το αντίστοιχο του παιχνιδιού με τον αμόλαφο που θα πρέπει να ε, κρίνουμε ποιος ε, θα ανέλθει στην ε, κορυφή και με ποια διαδικασία. Δεν πρέπει να θεσπίσουμε απαγορευτικά στοιχεία, σίγουρα να αποφεύγουμε τις καταχρήσεις, τις καταχρηστικές δηλαδή πρακτικές, αλλά θα πρέπει να δούμε και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς λειτουργούν τα κόμματα για να λειτουργούν αποτελεσματικά και να κερδίζουν τις εκλογές. Θα πρέπει να έχουμε ένα κλιμακωτό σύστημα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ε, έχουμε μια ε, εκπροσώπηση σε 13 χώρες και να αναγνωριστούμε ως κόμμα στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να μπορούμε να ε, αποδεικνύουμε ότι στις ευρωεκλογές έλαβα αυτό το ποσοστό. Και ε, με βάση αυτά τα στοιχεία να υπάρχει αποζημίωση για το κόστος της δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας. Διότι ε, ε, για να εκλεγεί κάποιος δεν θα πρέπει να ε, ξεπουλάει τα πάντα τα περιουσιακά του στοιχεία για να εξασφαλίσει μία θέση στην Ευρωβουλή. Επίσης θα πρέπει να δούμε την σχέση που υπάρχει μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, Περιφερειακών και της Ευρωβουλής. Ε, καλό είναι να καταργηθούν οι τεχνητές διαφορές. Για τα οικονομικά θέματα πρέπει να προσέξουμε κάτι ακόμα και το βλέπω και στις εργασίες του Προεδρείου του Κοινοβουλίου. Ε, υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που αφορούν ας πούμε, την αποφυγή του προσωπικού πλωτισμού. Ε, αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εμπόδιο αν ένα κόμμα πει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι τόσο σημαντικά ώστε να ε, με κάνουν να παρουσιαστώ με στεναρό τρόπο και να επηρεάσω την κοινή γνώμη. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και να αναγνωρίζεται. Θα πρέπει δηλαδή να, ε, όταν υπάρχει ε, θέμα σημαντικού πολιτικού στόχου θα πρέπει δηλαδή να μπορεί να ε, δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο ο βουλευτής και να μην αμφισβητούμε τα κονδύλια που τον έστειλαν στη Βαλένθια ή στο Ηράκλειο ή οπουδήποτε αλλού για να κάνει πολιτικές δηλώσεις και να έχει μια πολιτική παρουσία. Ε, είναι σημαντικό να μην ε, δρούμε ευνουχιστικά στα πολιτικά κόμματα. Τέλος, για την ατομική ιδιότητα του μέλους. Εγώ εδώ έχω μάλλον ευέλικτη στάση. Το 1984 σε ένα συνέδριο έγινε επίτιμο μέλος του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας. Γνωρίζω ανθρώπους που λένε εγώ θα αποχωρήσω διότι δεν συμφωνώ με τον επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης ε, και ή θα ήθελα να δραστηριοποιηθώ στο ανώτερο επίπεδο. Ε, βέβαια, ε, θα πρέπει να πούμε σε αυτούς ε, ότι δεν μπορεί κανείς να παρετηθεί ή να φύγει από την Εκκλησία επειδή δεν συμφωνεί με τον Πάπα. Ε, υπάρχουν, ε, η κυρία Γιαννάκου είπε πολλά σημαντικά. Αν ας πούμε ένα Ευρωπαϊκό Κόμμα δεν έχει πολιτική εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο. το Ευρωπαϊκό αυτό κόμμα για τη χώρα αυτή μπορεί να έχει να διαμορφώσει κάποιες ρίζες αν θέλετε, εν κενό και να πει ότι ο Πορτογάλος, παρόλο που ζει στις Βρυξέλλες και θέλει να γίνει μέλος, θα δημιουργήσω γι' αυτό το σκοπό μία ε, βάση για τη λειτουργία ε, του σε, αυτό το χώρο, σε αυτή τη χώρα. Ε, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης από εκλεγμένους βουλευτές και αν κάποιος ε, θέλει να ε, ενταχθεί σε ένα κόμμα, μπορεί να δημιουργηθεί εικονικά μια ε, ε, οργάνωση κόμματος και να υπάρχει έτσι η κομματική εκπροσώπηση. Δηλαδή ευέλικτες λύσεις υπάρχουν. Δεν θα μπορέσουμε να συνδυάζουμε λύσεις παράδοξες, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να ε, φτιάξουμε ένα αεροπλάνο που θα πετάει όταν έχει φτερό από τη μία πλευρά και τροχό από την άλλη. Ε, κύριε Γιαννάκου, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολλά σημαντικά και πράγματι ε, και όλοι οι ομιλητές προσπάθησαν να φύγουν και από τα στενά όρια ενός καταστατικού για ευρωπαϊκά κόμματα. Ε, τη δημιουργία ενός στάτους για τα ευρωπαϊκά κόμματα που στην ουσία προβλέπεται ήδη και από τον κανονισμό του 2003 ε, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το πρώτο βήμα. Το στάτους αυτό οφείλει να είναι πολιτικό καταρχήν, διότι η υπόθεσή μας είναι αμυγός πολιτική. Συνδέεται με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι πολίτες της Ευρώπης ε, τα ευρωπαϊκά πράγματα με την ανησυχία μας το είπε ο κύριος Γκερέρο πόσοι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές εκλογές στη χώρα μου κάποτε συμμετείχε το 95% και τώρα έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά το ποσοστό και στις ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και στις περιφερειακές εκλογές. Εάν λοιπόν τα κόμματα αυτά με πολιτικό τρόπο όπως τα αντιλαμβανόμεθα θέλουμε να μας βοηθήσουν με ένα καθεστώς και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο και νέο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά πράγματα στους πολίτες της Ευρώπης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το κυρίως πολιτικό θέμα. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό συμφωνώ και εγώ ότι ο ανταγωνισμός έχει σημασία διότι στη δημοκρατία η διαφωνία είναι πιο σημαντική τις περισσότερες φορές παρά η συμφωνία. Το δεύτερο ζήτημα είναι το δημοσιονομικό. Ποια κόμματα χρηματοδοτούμε. Δηλαδή μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα κόμμα που έγινε προχθές και δεν έχει καμία εκπροσώπηση είτε σε εθνικά κοινοβούλια σε ένα συγκεκριμένο αριθμό είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω κύριε συνάδελφοι ότι δεν μπορούμε. Πρέπει να αρχίσουμε με πολύ συγκεκριμένους τρόπους και με καλές πρακτικές ώστε τα επόμενα βήματά μας να έχουν θετικό πρόσημο. Να μην δημιουργηθούν δηλαδή αρνητικά στοιχεία τέτοια που δεν θα μας επιτρέψουν ούτε στους λαούς να κάνουμε γνωστές αυτές τις κινήσεις μας ούτε και σε επίπεδο <coughs> στελεχών ε, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων στελεχών στα διάφορα θεσμικά όργανα να μας κάνουν σεβαστούς. Ε, το τρίτο είναι το ε, φορολογικό σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα στάτους ευρωπαϊκού κόμματος που θα είναι σεβαστό το στάτους αυτό από όλα τα κράτη-μέλη, θα αναγνωρίζεται δηλαδή από όλα τα κράτη-μέλη, δεν θα υπερβαίνει τη συνθήκη, συμφωνώ με τον κύριο Βίλαντ, δεν είναι δυνατόν ακόμα αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε ότι μπορεί να εκλέγεται ο πρόεδρος της Επιτροπής, διότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, η Επιτροπή είναι εκτελεστική εξουσία. Το Συμβούλιο σε επίπεδο Ευρώπης είναι στην ουσία νομοθετική εξουσία αλλά ο διακυβερνητικός χαρακτήρας του συστήματος δεν έχει εγκαταληφθεί τελείως, ούτε έχει καταργηθεί και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν είτε να απαιτούμε να είναι ευρωβουλευτής ο Επίτροπος είτε να θέλουμε να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής διότι αν τον εκλέξουν οι λαοί τότε είναι υπέρτερος των συμβουλίων που αποφασίζουν και των αρχηγών κρατών που αποφασίζουν και είναι υπέρτερος από κάθε έλεγχο που μπορεί να το ασκηθεί από το Κοινοβούλιο ε, ή ε, άλλα, άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και επομένως νομίζω ότι το πρώτο βήμα μας πρέπει να είναι σταθερό και ολοκληρωμένο. Χρειαζόμαστε να περιβληθεί η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και όλα τα κόμματα είπαν ότι δεν χρειάζονται περισσότερα χρήματα ε, οι φιλελεύθεροι τόνισαν ότι πιθανόν να χρειάζονται περισσότερα. Αλλά δεν είναι το αντικείμενό μας αυτό. Νομίζω ότι ε, σε αυτό το σημείο θα έπρεπε ίσως να μας απαντήσουν με ένα ναι ή με ένα όχι συμμετέχοντες στη συζήτηση. Το πρώτο ολοκληρωμένο βήμα, χωρίς να αλλάξουμε τη συνθήκη, είναι η δημιουργία ενός στάτους πολιτικού, δημοσιονομικού και φορολογικού για τα κόμματα, τα ιδρύματά τους, τις νεολαίες τους και το staff των κομμάτων ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο που θα επιτρέψει εν συνεχεία όχι μόνο την ένταξη των κομμάτων αλλά και βεβαίως όπως όλοι είπαν ε, και την ένταξη μεμονωμένων προσώπων τα οποία θα μπορούν να γίνουν μέλη των κομμάτων αυτών. Θέλω να σημειώσω κύριε συνάδελφοι ότι επειδή υπάρχει διαφορετικό νομικό καθεστώς στις διάφορες χώρες θέλω να, να σας πω ε, ένα παλιό θέμα το οποίο όμως έχει σημασία. Κάποτε το κόμμα στο οποίο ανήκω εγώ θέλησε να δημιουργήσει όπως έκαναν και τα άλλα κόμματα στη Γερμανία οργανώσεις στο εξωτερικό. Συμβουλευθήκαμε νομικούς συμβούλους στη Γερμανία και μας είπαν ότι δεν μπορείτε να φτιάξετε κόμματα στη Γερμανία. Απαγορεύεται. Και μάλιστα το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην πατρίδα μας το είχε δημιουργήσει και δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα και απαγορεύτηκαν. Αν θέλετε μπορείτε να δημιουργήσετε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέγεται το κόμμα μας, ώστε να μπορείτε να είστε μέσα στη συνταγματική τάξη της Γερμανίας. Επομένως, επειδή έχουμε μεγάλες διαφοροποίησεις και επειδή και στη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Παραδείγματο χάρη στη χώρα μου χρηματοδοτήσει από το κράτος αν έχει εκπροσώπηση το Εθνικό Κοινοβούλιο ή αν έχεις τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εθνική δηλαδή χρηματοδότηση. Πόσο μάλλον η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει ανάγκη να υπάρχει εκπροσώπηση ε, στο κοινοβούλιο μας το οποίο εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και εκφράζει με τον ισχυρότερο τρόπο την ευρωπαϊκή δημοκρατία διότι το κοινοβούλιο την εκφράζει αυτή. Ήθελα λοιπόν να μας πούν έτσι με ένα ναι ή με ένα όχι οι αξιότιμοι κύριοι καθηγητές που πραγματικά μας έδωσαν ενδιαφέροντα στοιχεία αν αυτό είναι το σωστό και ολοκληρωμένο βήμα που πρέπει να κάνουμε τώρα. Το τι θα κάνουμε στο μέλλον και πώς εξελίσσονται τα πράγματα ξέρουμε ότι στην Ευρώπη συνεχώς εξελίσσονται. Δεν σταματούν ποτέ και δεν θα σταματήσουν κατά τη γνώμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από αυτό. Λοιπόν, ρωτώ του τρει ε, εμπειρογνωμονε μα, ε, αν θέλουν ε, να αντιδράσουν στις ερωτήσεις ή στι προκλήσεις των μελών. Για να μπορέσουμε όμως να κρατήσουμε το χρόνο μας, επειδή έχουμε να ακούσουμε κι άλλους, μόνο τρία λεπτά ο καθένας, αλλά σε τρία λεπτά Προλαβαίνει να πει κάτι κανείς. Να πάμε με τη σειρά. Ο καθηγητής Μόρλοκ θέλει το λόγο. Ο κύριος Χέφνερ έκανε τρεις ερωτήσεις από ό,τι κατάλαβα. Πρώτον, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να ε, χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό τα ευρωπαϊκά κόμματα. Δεν έχω σίγουρη απάντηση, Πάντως δεν θα πρέπει να είναι η προϋπόθεση η ένταξη στο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ ψηλό το εμπόδιο. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Επίσης τα κόμματα δεν είναι, ε, είναι εκπρόσωποι των πολιτών, δεν είναι μόνο ε, τμήματα του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, να λειτουργούν τα κόμματα και να τα βλέπουμε μέσα από αυτό το πρίσμα. Ε, κόμματα που εκπροσωπούνται σε πολλές χώρες, που έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό δεν θα ήθελα να πω, αλλά το Συνταγματικό Δικαστήριο στη Γερμανία πριν από λίγα χρόνια ε, αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγματική μία διάταξη ότι θα χρηματοδοτούνται τα κόμματα μόνο αν ε, εκπροσωπούνται ε, με 1% τουλάχιστον σε 3 από 16 ε, κρατήδια. Ε, αυτό θεωρήθηκε συνταγματικό. Πρέπει λοιπόν να μην είναι πολύ ε, υψηλά τα εμπόδια που βάζουμε, διότι χρηματοδοτούνται ε, επειδή συγκεντρώνουν ψήφου από πολίτε στα κόμματα. Τώρα για την εσωκομματική δημοκρατία, εκεί χρειάζονται κανόνες και έμαθα από τον κύριο Μπάρντι ότι η απάντησή μου ε, δεν ήταν λίγο βεβιασμένη. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι ιδιαίτερα οργανισμοί και θα πρέπει ίσως να προβλέψουμε ε, κάποια χαλαρά ε, συστήματα, χαλαρότερα τουλάχιστον. Εδώ χρειάζεται να είμαστε εφάνταστοι. Ε, παρόμοια θα έλεγα και για το τρίτο θέμα, την ατομική και συλλογική ιδιότητα του μέλους παράλληλα. Αυτά δεν είναι μόνο ανεπίλητα προβλήματα, αλλά προβλήματα τα οποία, πάνω στα οποία δεν έχουμε παρκώς ε, στοχαστεί. Ε, Επίση, για την ερώτηση της κυρίας Γιαννάκου, η Νέα Δημοκρατία στη Γερμανία δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, διότι το δίκαιο για, τις, για τα κόμματα ε, περιορίζεται στην εθνική ε, προοπτική. Ε, γι' αυτό χρειάζεται μια ευρωπαϊκή ε, νομική μορφή για τα πολιτικά κόμματα. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής Μπάρντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα απαντήσω πολύ σύντομα στις τρεις ερωτήσεις. Πρώτο, κριτήρια. Για να είναι κανείς Ευρωπαϊκό Κόμμα. Είπα σαφώς ποια ήταν η θέση που υποστηρίζω για τα πολιτικά κόμματα και την, αντιπροσω... την εκπροσώπησή τους. Αυτή ήταν και γνώμη των υπολείπων συναδέλφων του παρατηρίου. Υπό το φως των όσων είπαν και άλλοι, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται για τους λόγους που ανέφερε και ο κύριος Μόρλοκ η εκλογή του ενός μέλου στο Κοινοβούλιο. Είναι πολιτική η λύση και η απόφαση και αυτό εμπίπτει σε αυτούς που ασκούν την πολιτική ως επάγγελμα και όχι σε μας. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι αυτή η περαιτέρω σκλήρινση δεν είναι απαραίτητη για την εσωτερική δημοκρατία. Ναι, Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, εμείς αναφέραμε μερικούς που ήδη σε εθνικό επίπεδο έχουν μια ανταπόκριση. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο το οποίο πρέπει να επικυρώσουμε. Εσωτερικές εκλογές, ένας πρώτος γύρος δυνατότητα ατομική membership. Νομίζω ότι απάντησα σαφώς στο ναι ή όχι της εισηγήτριας ότι το κριτήριο του εκλεγμένου μέλου στο κόμμα δεν είναι απαραίτητο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένας διαχωρισμός μεταξύ της έννοιας του τι αποτελεί ένα ευρωπαϊκό κόμμα και το δικαίωμά του για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση δίνεται στην φάση ανάπτυξης των κομμάτων. Το να μην χρηματοδοτούνται τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στο κοινοβούλιο θα ήταν πραγματικά ε, μία τροχοπέδηση της δυνατότητας ανάπτυξης του δίου του κόμματος. Το, το άλλο θέμα είναι πάρα πολύ ευρύ για να το συζητήσουμε εδώ. Καθηγητής Χρυσοχώου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αναλύσω λεπτομερώς αυτά που συζητήσαμε για τις προτινόμενες αλλαγές. Θα απαντήσω μόνο καταφατικά στην ερώτηση της κυρίας Γιαννάκου και θα πω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια σταδιακή προσέγγιση αυξητική λόγω της φύσης της και όχι μια βεβαιασμένη προσέγγιση που πάει να ε, επιτύχει μαξιμαλιστικούς στόχους. Ε, που δεν θα μπορέσει να αφομοιώσει και να εναρμονίσει στα πλαίσια της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αναγνώρισης θα έλεγα ότι ναι είναι δυνατόν όπως είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο να υπάρξει πιθανώς μια χαλάρωση των κριτηρίων και αυτό να είναι θετικό αλλά πρέπει να είμαστε σταθεροί σχετικά με το αν τα ευρωπαϊκά αυτά κόμματα χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να έχουν εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι εδώ η απάντηση είναι σαφής. Εγώ συμφωνώ με την έκθεση. Σύμφωνο με την ευρύτερη συνένεση που φαίνεται να ε, διαμορφώνεται ότι θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένα μέλος εκλεγμένο στο Ευρωκοινοβούλιο. Για την ε, ιδιότητα του μέλους που είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε στη συζήτηση και εδώ αρχίζει να διαμορφώνω μια άποψη, εδώ κατά τη συζήτηση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να, να ψάξουμε να βρούμε τρόπους ε, εισαγωγής ε, της έννοιας ε, της ατομικής ιδιότητας του μέλους. Μπορεί να μην είναι από νομικής άποψης τόσο εύκολο όσο φαντάζεται κανείς με την πρώτη ματιά. Αλλά το να ε, χορηγήσει κανείς ένα καθεστώς υποστηρικτή οπαδού μπορεί να μην επαρκεί για να προκαλέσει ή να κινητροδοτήσει ή να κινητοποιήσει τα ε, ουσιαστικά αυτά στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη. Μπορεί λοιπόν, θα έλεγα, να χρειάζεται να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο και μπορεί ίσως να υπάρξει και μια υβριδική φόρμουλα, κάτι μεταξύ ιδιότητας μέλους ή οπαδού ή μια πιο χαλαρή μορφή ιδιότητας μέλους, αλλά η ιδιότητα του μέλους νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για να ε, δράσει καταλυτικά και να δημιουργήσει μια ταύτιση, ταυτοποίηση. Ευχαριστώ συλλογικά όλους τους εμπειρογνώμονες. Πάμε στο επόμενο σημείο. Ο δόκτωρ Λουίς Γκαλέα, ο οποίος είναι μέλος του Ερεκτικού Συνεδρίου και θα μας δώσει τη δική του ανάλυση για τα χρημα... τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις σημερινές συζητήσεις που ήταν πραγματικά συναρπαστικές γιατί έβριθαν εύστοχων σημείων και πραγματικά συναρπαστικών και φάνταστων ιδεών. Ε, βέβαια, ο ρόλος του ε, ελεκτικού συνεδρίου είναι κάπως πιο νοσηρός ε, είναι πιο μακάβριος και θα ήθελα εκ των προτέρων να ζητήσω συγγνώμη για αυτού του είδους ε, τις πένθυμες και νοσηρές σκέψεις που θα σας εκθέσω. Όπως σας είπα, είμαι ε, εκπρόσωπος εδώ του Ελεκτικού Συνεδρίου και σας ευχαριστώ θερμά που προσκαλέσατε και το Ελεκτικό Συνέδριο για να εκφέρει τις θέσεις τους ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, κομμάτων. Βέβαια αυτή είναι πιο πεζή προσέγγιση ε, σε σχέση με τα προηγούμενα εφάνταστα σχόλια που ακούσαμε. Αλλά θα προσπαθήσω να σας εκθέσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις σκέψεις. Τέτοια κόμματα είναι επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση από το κοινοτικό προϋπολογισμό με τη μορφή επιδοτήσεων που μπορεί να χορηγηθούν από το, να χορηγηθούν από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στο πλαίσιο αυτό είναι ένα κεντρικός ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου, ο ρόλος ε, του ελέγχου, της παρακολούθησης και της ε, ενημέρωσης ε, σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και επίσης να εκφέρει γνώμη σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά για το κατά πόσο είναι συμβατή αυτή η χρήση με τη συνθήκη. Δεν είμαι σε θέση σήμερα να σας υποβάλω την επίσημη θέση του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά θα σας δώσω κάποιες γενικές σκέψεις για το πλαίσιο και τους βασικούς προσανατολισμούς της συζήτησης και της διαμόρφωσης σκέψης μας. ό,τι αφορά την εκτίμηση, την αξιολόγηση για τη χρηματοδότηση και την δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα υπό τρεις πτυχές. Καταρχήν, η πρώτη πτυχή είναι η ερμηνεία των απαιτήσεων της συνθήκης. Η δεύτερη είναι οι κανόνες του κανονισμού 2004-03 σε συνδυασμό με τους εφαρμοστικούς κανόνες και τρίτο θέμα, τρίτη πτυχή είναι η συμμόρφωση με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών μέτρων. Θα αναφερθώ στις πτυχές αυτές ξεχωριστά. Ε, οι διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 4 της Συνθήκης, ε, προβλέπουν την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ευαισθητοποίησης και της έκφρασης ε, της βούλησης των πολιτών και επίση περιλαμβάνουν την έννοια ότι τα, τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμβάλλουν σημαντικά στην ε, ενίσχυση αυτών των θεμάτων. Επίσης, η συνθήκη χρησιμοποιεί τον όρο πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αυτό προϋποθέτει την ανάγκη ενός ορισμού που θα υπερβαίνει το απλό γεγονός ότι ένα πολιτικό κόμμα προέρχεται από ένα μονοκράτος μέλος, αλλά απαιτεί μια προοπτική που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Σε μια ένωση που απαρτίζεται από κράτη-μέλη, αναμένεται ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα τα πολιτικά κόμματα, θα έχουν τις ρίζες τους σε μεμονωμένες χώρες. Παρ' όλα αυτά, η συνθήκη δεν φαίνεται να ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στην δυνητική δυνάμη, μάλλον προς τη θέμενη αξία, δηλαδή την προαγωγή των δημοκρατικών ιδεωδών και πρακτικών στην Ένωση, ε, έχοντας ε, τα πολιτικά κόμματα που υιοθετούν μια ευρύτερη πανευρωπαϊκή προοπτική. Το προήμιο του κανονισμού 2004-03 προβλέπει στην παράγραφο 4 το εξής ε, κριτήριο. Προκειμένου να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να θεσπίσουμε κάποιες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερα είναι απαραίτητο τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τηρούν τις αρχές, να σέβονται τις αρχές στις οποίες ε, στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κατοχυρώνονται από τις συνθήκες και αναγνωρίζονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός αυτός, στα άρθρα 2 και 3, παρουσιάζει έναν ορισμό των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβάνοντας και μια σειρά προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται. Στις ε, αν οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες του ορισμού αυτού θα υποστούν αναθεώρηση, οι προτινόμενες τροπολογίες θα πρέπει να σέβονται τις διατάξεις της συνθήκης ή τα κριτήρια της συνθήκης. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομεριακέ παραθέσει. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο κανονισμό 2004-03 καλύπτει και τα πολιτικά ιδρύματα εκτό από τα πολιτικά κόμματα. Και ο ορισμό του, του πρώτου όρου των πολιτικών ιδρυμάτων συσχετίζεται με το δεύτερο όρο, τα πολιτικά κόμματα δηλαδή. Επίσης, πέραν των προναφερθησών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται από τα κόμματα, ο κανονισμός ε, προβλέπει μεταξύ άλλων ποιοι θα είναι οι εφαρμοστέοι κανόνες ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση, προσδιορίζει τις ε, τη χρήση των κονδυλίων και επίσης ε, προβλέπει τον τρόπο καταμερισμού των διαθέσιμων κονδυλίων και πιστώσεων. Και πάλι θα αποφύγω την λεπτομεριακή παράθεση των άρθρων 6, 7, 8 και 10 του κανονισμού που προσδιορίζουν ακριβώς με περισσότερες λεπτομέρειες αυτά τα σημεία. Πριν την διοργάνωση αυτής της ακρόασης, η συγγήτρια μας είχε υποβάλει ένα ερωτηματολόγιο με πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να ανακύψουν στη διάρκεια της συζήτησης. Μερικές ερωτήσεις αφορούν τη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, τα κριτήρια της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης που προβλέπει ο κανονισμός είναι υπερβολικά αυστηρά ή υπερβολικά γενναιόδωρα. Το κλειδί για, την κατα... για τον καταμερισμό των διαθέσιμων πιστώσεων είναι ο πιο ορθολογικός. Είναι ε, κατάλληλο το κριτήριο της αυτοχρηματοδότησης. Είναι αναφυσβήτητο ότι τα πολιτικά κόμματα αποτελούν ζωτικό εργαλείο και απαραίτητο για την εύρυθμη εφαρμογή ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος. Οπότε οποιαδήποτε διεύρυνση των, δραστηριοτήτων θα ήταν ευπρόσδεκτη. Βέβαια και είναι πιθανές οι αλλαγές, θα πρέπει να εξεταστούν και επίσης οι εφαρμοστικοί κανονισμοί θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις ε, με τα κριτήρια των κανονισμών και αυτών συντακτών τους. Στον έλεγχο της νομιμότητας ε, και τακτικότητας, το ελεκτικό συνέδριο θα εξετάσει σε ποιο βαθμό ε, υπήρξε συμμόρφωση με τους κανόνες και το κατά πόσο οι προβλεπόμενοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν για τους υλοποίησεις σκοπών που είχαν προσδιοριστεί. θα πρέπει να δούμε αν υπήρξε περιορισμό στο κονδυλίο ή περιορισμό τη αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων. Βέβαια, υπερβολικέ λεπτομέρειε και μία πληθώρα εξαιρέσεων ίσω ε, ε, δυσχεράνει τη λειτουργία του χρηματοδοτικού κανονισμού. Σε πολλέ περιπτώσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρονομοδότηση για δημοσιονομικό κανονισμό και για παρόμοια εργαλεία, το ελεκτικό συνέδριο έχει τονίσει ότι οι περίπλοκοι κανόνες ή ασαφή κριτήρια επιλεξιμότητας έχουν ε, ε, σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ομιμότητα και την τακτικότητα των ε, συναλλαγών. Και επιπλέον, μια περίπλοκη διάταξη αυξάνει το κόστος της συμμόρφωσης και του ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τώρα την επαλήθευση και τα ελεκτικά μέτρα. Είναι αυτονόητο ότι τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να χαίρουν της απαραίτητης ελευθερίας προκειμένου να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους ε, εν πλήρη ανεξαρτησία. Οι, οι διάφορες δομές ε, που διέπουν την διαχείριση των δημοσίων κονδυλίων των πολιτικών κομμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την ελευθερία τους επουδενή. Βέβαια, τα ελεκτικά μέτρα, χρειάζονται κάποια ελεκτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι πιστώσεις καταβάλλονται και χρησιμοποιούνται ε, με βάση τον κανονισμό και για τους σκοπούς που προσδιορίσε ο νομοθέτης. Οι κανονισμοί δεν θα είναι αποτελεσματικοί αν δεν συνοδεύονται από αποτελεσματικά ελεκτικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη σωστή συμμόρφωση με τον κανονισμό. Και αυτό είναι ένας άλλος παράγοντας που χρήζεται διεξοδική ανάλυση. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό ε, η χρηματοδότηση και η δημοσιονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνοδεύεται από διατάξεις για ένα κατάλληλο ελεκτικό πλαίσιο. Το άρθρο 5 του κανονισμού αναφέρει ρητά την ανάγκη για συνεχή επαλήθευση και έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των όρων υπό τους οποίους χρηματοδοτούνται τα κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο ενός αποτελεσματικού ελεκτικού συστήματος. Γιατί η έλεγχη είναι ένα τμήμα της λειτουργίας του συνολικού συστήματος. Το άρθρο 9 αναπτύσσει περαιτέρω το θέμα του ελέγχου. Γιατί είναι γενική αρχή ότι ο έλεγχος των κονδυλίων που προβλέπονται από τον κανονισμό θα ασκείται με βάση τον δημοσιονομικό κανονισμό και τις εφαρμοστικές του διαδικασίες. Η αρχή αυτή θα πρέπει να διαφυλαχθεί και καμία τροποποίηση του κανονισμού 2004-03 δεν θα πρέπει να προταθούν αν δεν ευθυγραμμίζονται με το δημοσιονομικό κανονισμό, εκτός και αν θεωρείται κάτι τέτοιο πιθανό και δικαιολογημένο να τροποποιηθεί και ο δημοσιονομικός κανονισμός. Θα σας υπενθυμίσω την κατάσταση που είχαμε το 2007 με την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού. Τότε η σε σχέση με τις επιδοτήσεις, οι εξαιρέσεις από τον μη κερδοσκοπικό κανόνα του δημοσιονομικού κανονισμού είχε θεσπιστεί υπέρ των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο άρθρο 109 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπεται ότι οι επιδοτήσεις δεν πρέπει να έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την προσκόμιση ωφέλους για τον δικαιούχο. Βέβαια υπάρχει και εξαίρεση από τον κανόνα αυτό που προβλέπει ότι είναι ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιεί πλεόνασμα εισοδήματο ε, από τον δαπανών για το, προς το τέλος του, της δημοσιονομικής χρήσης, ένα τμήμα αυτού του πλεονάσματος μέχρι 25% του συνολικού ε, εισοδήματο του έτους μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο έτος, αρκεί να χρησιμοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, του επόμενου διαχειριστικού έτους. Τότε μάλιστα το, Ευρωπαϊκό, το Ελεκτικό Συνέδριο είχε δώσει τη γνώμη 7-2007 και ένα από τα συμπεράσματα αυτής της γνωμοδότησης ήταν ότι οι σαφείς ορισμοί των όρων ε, δημοσιονομικά αποθέματα και μέσω ετήσιο εισόδημα ήταν απαραίτητα για να δικαιολογηθεί η σωστή εφαρμογή και επαλήθευση του, των εξαιρέσεων από τον μη κερδοσκοπικό κανόνα. Δυστυχώ, οι συστάσει τη γνωμοδότηση δεν ε, ελήφθησαν υπόψη και δεν έγιναν περαιτέρω τροποποίηση στο, στο δημοσιονομικό κανονισμό. Παρόλο που προβλέπεται ότι ο έλεγχος θα ασκείται επί τη βάση της αιτήσεως πιστοποίησης από έναν ανεξάρτητο και εξωτερικό ελεκτή, η χορήγηση επιδοτήσεων από το κοινοτικό προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα υπόκειται στον έλεγχο του εσωτερικού ελεκτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, που είναι ο εξωτερικό ελεκτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλο του Ελεκτικού Συνεδρίου καλύπτεται ρητά στον κανονισμό 2004-03 που προβλέπει ότι οποιαδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που θα απαιτείται από το ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να διενεργήσει το, την αποστολή του θα πρέπει να υποβάλλεται κατά από τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφόσον λαμβάνουν επιδότηση με βάση τον κανονισμό. Και όταν ε, κάποια δαπάνη γίνεται από πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από κοινού με εθνικά κόμματα ή άλλες οργανώσεις, η απόδειξη των δαπανών των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προσκομίζεται στο ελεκτικό συνέδριο. Η πρόσβαση του ελεκτικού συνεδρίου σε έγγραφα που αφορούν χρηματοδότηση της, του ευρωπαϊκού προπολογισμού κατοχυρώνεται και περιχαρακώνεται στο άρθρο 289, παράγραφος 3 της συνθήκης. Παρ' αυτά, το το δικαίωμα πρόσβασης αυτής αναφέρεται ρητά και στον κανονισμό που αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και οι σχετικές παράγραφοι θα πρέπει να τηρηθούν και να διαφυλαχθούν. Θα σας πω δύο λόγια και για τις προοπτικές του ελεκτικού συνεδρίου. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο είναι το ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που έχει θεσπιστεί από τη συνθήκη για να διενεργεί τον έλεγχο των ευρωπαϊκών οικονομικών λογαριασμών μια και είναι εξωτερικό ελεκτή, το ελεκτικό συνέδριο είναι ανεξάρτητο από τα άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελέγχει τη σωστή λογιστική απόδοση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και την χρησιμοποίησή του ε, με βάση του κοινοτικού κανόνε και νομοθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη αξιοποίησή του. Επίση, το ελεκτικό συνέδριο τηρεί τι διεθνεί προδιαγραφέ ελέγχου όπως εφαρμόζονται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Προκειμένου να εξασφαλίσει την ε, συμμόρφωση του τρόπου ε, δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ε, ε με, με τις διάφορους κανονισμούς και το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να κάνει σωστή ε, εξέταση από τα εποπτικά και ελεκτικά όργανα και να εντοπίσει πιθανά λάθη και ατασταλίες σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές. Και μάλιστα τα αποτελέσματα του, ε, του ετήσιου ελέγχου της, του ελεκτικού συνεδρίου δημοσιεύονται ετησίως με τη μορφή ε, δήλωσης ε, που είναι γνωστή ως DAS, δήλωση αξιοπιστίας, που είναι γνωστή ως DAS. Σε ό,τι αφορά την ε, διενέργεια του ελέγχου, το δικαστήριο έχει μια σειρά ελεκτικών μεθοδολογιών με βάση τα κριτήρια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών ε, δημοσιεύονται και σε ειδικέ εκθέσεις. Ακόμη και στη αν στη διάρκεια των ελέγχων το ελεκτικό συνέδριο εντοπίσει τα σταλίες που δημιουργούν υπόνοιες για απάτη, μπορεί να υποβάλει αναφορά στην ειδική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη της απάτης και της διαφθοράς, την ΟΛΑΦ. Σε ό,τι αφορά τις ε, χρηματοδοτήσεις και τις πιστώσεις των πολιτικών κομμάτων, οι δαπάνες αυτές καλύπτονται στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας της, του ελεκτικού συνεδρίου, μαζί με τα άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν τμήμα της Γενικής Ομάδας Πολιτικής που φέρει τον τίτλο «Διοικητικές δαπάνες». Μέχρι στιγμής ε, το Ελεκτικό Συνέδριο ουδέποτε δεν ασχολήθηκε μόνο με τον έλεγχο της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο μέλλον όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και στόχος μας είναι να εκδώσουμε ειδική έκθεση για το θέμα αυτό. Ένα σημαντικό τμήμα τέτοιου ελέγχου θα είναι μία εκτενής αξιολόγηση του κινδύνου προκειμένου να εντοπίσουμε τους πιθανούς κινδύνους και απειλές στην ε, τακτικότητα και την ομιμότητα των ε, ροών ταπανών σε συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν ε, μερικά παραδείγματα δυνητικών κινδύνων που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και να αναπτυχθούν στα πλαίσια μίας κανονικής ανάλυσης των επιπτώσεων. Πιθανές, πιθανή κίνδυνη μία νομική οντότητα ε, μπορεί να έχει δεχτεί τα κονδύλια χωρίς να πληρεί τις ε, προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν τηρεί ή αθετεί κάποιες υποχρεώσεις. Μία αίτηση μπορεί να έχει γίνει δεκτή με ανακριβή ή ε, μη πλήρη στοιχεία. Η χρηματοδότηση μπορεί να δίνεται για στόχους διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει ο κανονισμός ή μπορεί να δίνεται σε οντότητες που παραβιάζουν τους κανονισμούς οι πιστώσεις, μπορεί, οι δαπάνες μπορούν να μην έχουν ε, αναφερθεί σωστά ή να μην συνοδεύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Η εξωτερική πιστοποίηση μπορεί να μην καλύπτει επαρκώς όλα τα πετούμενα κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετριαστούν αισθητά οι προαναφερθέντες κίνδυνοι, που είναι η διοικητικές ε, ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωση με τους κανόνες. Βέβαια, περαιτέρω ανάλυση του θέματος αυτού είναι απαραίτητη. Αλλά η δυνατότητα επιβολή τέτοιων ε, διοικητικών κυρώσεων προβλέπεται ήδη στον κανονισμό 2988 κάθετο 95 της 18 Δεκεμβρίου του 1995 του Συμβουλίου με θέμα την προστασία των ε, χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τελευταίο σημείο είναι η διαφάνεια. Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε υπόψη τις διατάξεις το, της αιτιολογικής έκθεσης του κανονισμού 2004-03 που προβλέπουν ρητά και κατηγορηματικά ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια και δημοσιονομικός έλεγχος των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που χρηματοδοτούνται από το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός ε, απαιτεί συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημοσιεύσει μια σειρά εκθέσεων και επίσης έναν αιτήσιο, ε, έναν απολογισμό των ποσών και των επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε κάθε πολιτικό κόμμα και πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικέ οι διατάξει αυτέ και όπου δει θα πρέπει να ενισχύονται. Το 2003 το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη φορά, του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθέτησε τη σύσταση παριθμών 4 για κοινού κανόνε για πάταξη τη διαφο σε χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και προεκλογικών εκστρατείων. Η σύσταση αυτή αναφέρεται στην ανάγκη ε, αύξηση της διαφάνειας ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Και μάλιστα η εφαρμογή της σύστασης αυτής ελέγχεται από την ομάδα Γκρέκο, την ομάδα κρατών κατά της ε, διαφθοράς που ιδρύθηκε το 1909 από το Συμβούλιο της Ευρώπης προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση ε, με, τα, με τις προδιαγραφές πάταξης της διαφθοράς και μάλιστα το Μάιο του 2010 δημοσιεύθηκε μια συγκριτική ανάλυση σε 22 από τα 47 κράτη που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ίσως υπάρχει χάσμα μεταξύ του γράμματος του νόμου και της έμπρακτης εφαρμογής του. Η ανάλυση αυτή τόνισε την ανάγκη οποιαδήποτε αξιολόγηση της διαφάνειας χρηματοδότης πολιτικού κόμματος ε, ε, θα πρέπει να επικεντρώνεται στην συμμόρφωση του υπάρχοντος κανονισμού και της ανάγκης επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες αυτού του κανονισμού. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω ότι ο κανονισμός ε, περιέχει έναν ορισμό των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και περιλαμβάνει μια σειρά προϋποθέσεων που θα πρέπει να συντρέχουν. Αν οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες του ορισμού αυτού υποστούν ε, ε, τροποποίηση, οι προτινόμενες αλλαγές θα πρέπει να σέβονται τις διατάξεις της συνθήκης. Οι κανονισμοί μπορεί να τροποποιούνται με τη, με τη διαγραφή ενός τμήματων ή με την προσθήκη ε, λεπτομεριών εξαιρέσεων ε, ίσως η έλλειψη λεπτομέρειας δημιουργήσει μια συγκεχημένη κατάσταση, αλλά η πληθώρα λεπτομεριών ίσως ε, κάνει τον μηχανισμό πιο δύσχριστο. Είναι σημαντικό οι εφαρμοστικοί κανονισμοί να ευθυγραμμίζονται με το δημοσιονομικό κανονισμό. Καμία αλλαγή του κανονισμού 2004-03 δεν θα πρέπει να προτείνονται εφόσον αντιβαίνουν στο δημοσιονομικό κανονισμό, εκτός φυσικά και αν θεωρείται δυνατό και δικαιολογημένο να τροποποιηθεί και ο δημοσιονομικός κανονισμός. Η πρόσβαση του ελεκτικού συνεδρίου σε δικαιολογητικά και έγγραφα που αφορούν χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό περιχαρακώνεται στη συνθήκη. Επίση είναι σημαντικό το δικαίωμα πρόσβασης να αναφέρεται ρητά και στον κανονισμό 2004 και θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι λόγω παράγραφοι του κανονισμού 2004. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μετριαστούν οι κίνδυνοι μη τήρησης των κανόνων. Οι διατάξεις για την πρόθεση της διαφάνειας είναι πολύ σημαντικές και όπου δεν θα πρέπει να ενισχύονται. Το ελεκτικό συνέδριο, κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε στη δημόσια αυτή ακρόαση. Ε, μία ακρόαση που περιστράφηκε γύρω από τον τρόπο χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον και αν έχουμε συγκεκριμένε αλλαγέ στον κανονισμό 2004-03 αναμένεται διαβούλευση με το ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να δημοσιευθεί σχετική γνωμοδότηση το πνεύμα φυσικά του κοινού στόχου που είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Ευχαριστώ καθηγητά Γκάλερ για την πλήρη έκθεσή σας. Αναλυτικότατη. Ο κύριος Βίλαν ζήτησε να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκαλέα, πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Ε, κάτι σημαντικό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Πολλές φορές μιλάμε για κονδύλια με συγκεκριμένο σκοπό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Ε, αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μας απασχολήσει γιατί θα ήταν λάθος να πούμε ότι αν χρηματοδοτήσουμε ένα κόμμα μετά θα πρέπει να ελέγχουμε πού δαπάνησε ακριβώς τα κονδύλια αυτά το κόμμα. Υπάρχουν ρευστά όρια στα πολιτικά περιεχόμενα και εκεί νομίζω ότι πρέπει να κρατηθούμε κάπως μακριά. Από ό,τι γνωρίζω εγώ τη λειτουργία των κομμάτων και την πραγματικότητά τους στα κράτη-μέλη, ε, με βάση αυτά που γνωρίζω θα έλεγα ότι αν κάποιος χρηματο... χρησιμοποιήσει κονδύλια, ε, τότε το κόμμα θα πρέπει να φροντίσει να μην λείψουν τα κονδύλια αυτά. Δεν είναι η κορυφή του κόμματος που θα χρησιμοποιήσει τα κονδύλια και θα τα πάρει από το ταμείο του κόμματος πολλές φορές ε, ε, μεμονωμένοι ε, πολίτες ε, ε, κρατούν αποστάσεις από τα κόμματα για να εξασφαλίζουν καλύτερο έλεγχο. Εάν ε, προσχηματικά τα κόμματα ζητήσουν και αποκτήσουν κονδύλια, αυτό θα πρέπει να το τιμωρούμε, θα πρέπει να υπάρχουν δηλαδή κυρώσεις εδώ, αλλά αν ένα κόμμα νομοτύπος απέκτησε κάποια κονδύλια θα πρέπει να έχει κάποια ελευθερία χειρισμού γιατί πρέπει να υπάρχει και πολιτική ελευθερία των κομμάτων. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα πολυεπίπεδο σύστημα κοινοβουλευτισμού και ε, κομματικής λειτουργίας ε, παρεμβαίνοντας ε, αυθαίρετα σε επίπεδα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια ελευθερία για το που δόθηκαν για την ενίσχυση των, ε, της δομής του κόμματος ε, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να δρούμε αποτρεπτικά εκεί. Επίσης, ε, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί όπου οι πολιτικοί σχηματισμοί ε, χρηματοδοτήθηκαν σε ένα κοινοβούλιο, εκεί θα πρέπει να ισχύει ότι δεν θα πρέπει εκεί εμέσως να χρηματοδοτούνται τα κόμματα, ούτως ώστε εκείνοι που βρίσκονται στο κοινοβούλιο να βοηθούν νοθεύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των βουλευτών και των μη βουλευτών μελών ενός κόμματος. Πιστεύω ότι είναι λάθος ε, να αναγκάζονται τα κόμματα το 25% των ε, κονδυλίων τους να τα ε, ε, δαπανούν ε, το επόμενο έτος. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία στα κόμματα. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να πει δηλαδή το κόμμα ότι ε, κάθε χρόνο κρατάμε το 50% του προϋπολογισμού μας για να το δαπανίσουμε στις ευρωεκλογές. Αυτό θα πρέπει να είναι ε, δεδομένο για τα κόμματα. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα σχετικά με ε, νόμιμα αποκτηθέντα έσοδα. Θα πρέπει αυτό να επιτρέπεται. Επίσης, ε, το ελεγκτικό συνέδριο σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να σιωπά όπως το Μαντίο των Δελφών και εκ των υστέρων να υποβάλει παρατηρήσεις και σχόλια, θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο εκ των προτέρων να λέει ότι ναι, αυτές οι πρακτικές μπορεί να είναι θεμητές και πιστεύουμε ότι οι γενικοί κανόνες θα πρέπει να ισχύουν και να είναι αυτοί και όχι άλλοι. Ο κύριος Έφνερ. Μετά ε, θα μιλήσει η κυρία Μετερμάιερ. Παρόμοια ερώτηση θέλω να κάνω. Είναι σημαντικό το ελεγκτικό συνέδριο να εξετάζει πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα θέματα. Πολλές φορές όμως οι ρυθμίσεις μας είναι γραφειοκρατικές και περιοριστικές. Ενώ τώρα υπάρχει ευκαιρία να διορθώσουμε πολλά. Σας ερωτώ λοιπόν, η τωρινή πρακτική ποια είναι. Δεν υπάρχει ανάγκη εκ των προτέρων να ε, υποβάλουν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων τα κόμματα και αυτό καμιά φορά δεν περιορίζει την ελευθερία της ε, αντιπαράθεσης. Ίσως θα, καλύτερη θα ήταν μια άλλη ρύθμιση η οποία θα συνέδεε τη χρηματοδότηση των κομμάτων σε αντικειμενικούς παράγοντες που καθορίζονται από τους πολίτες, τους ψηφοφόρους και που θα διασφαλίζουν κάποια κονδύλια για το κόμμα ε, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία για τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων σε δημοκρατικά πλαίσια και σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Νομίζω ότι περιορίζεται έτσι η γραφειοκρατία και περιορίζεται ο έλεγχο σε σοβαρές περιπτώσεις. Δεν είναι χρήσιμο να απαιτούμε την επιστροφή των χρημάτων, αλλά όταν υπάρχουν καταχρήσεις, όπου υπάρχει παράβαση, παραβίαση της ε, νομοθεσίας, εκεί θα πρέπει να προβλέπονται αποτρεπτικά μέτρα, ούτως ώστε να αποτρέπονται στο μέλλον ε, τέτοιες πρακτικές. Αν θέλετε να απαντήσετε, πρέπει να ακούσουμε όμως και την κυρία Μίτερ Μάγερ για τη διαφάνεια. Υπάρχουν και άλλες τοποθετήσεις. Παρακαλώ λοιπόν τον καθηγητή Γκάλεα να απαντήσει σε αυτές τις τοποθετήσεις. Μετά θα μιλήσει η κυρία Μίτερ Μάγερ και μετά ζήτησε και ο κύριος Νταφ το λόγο. Θα μπορούσε ίσως στο τέλος να μιλήσει ο κύριος δαφ και να δούμε όλο το υλικό μαζί. Καθηγητής Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω σύντομα και στα δύο αξιότιμα μέλη. Σχετικά με το πρώτο θέμα του κυρίου Βίλαντ. Ναι, συμφωνούμε, έχει συμφωνηθεί, ότι η πόροι αναμένεται όχι μόνο να ε, χρησιμοποιούνται για τους συγκεκριμένους σκοπούς, ε, όχι μόνο να ανατίθενται για συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά να δαπανώνται για τους συγκεκριμένους σκοπούς και αυτό να αποδεικνύεται με βάση συγκεκριμένα τεκμήρια. Προλόγης, ε, στήριξα την παρέμβασή μου στην σημαντική αρχή της διασφάλισης της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των πολιτικών κομμάτων. Και αυτό ε, είναι ένα θέμα που έθιξαν πολλοί ε, συμμετέχοντες και ομιλητές. Το ελεγκτικό συνέδριο, το μόνο που υποχρεούται να κάνει, είναι να ελέγχει. Γι' αυτό η συνθήκη του δίδει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό είναι ο εξωτερικός έλεγχος. Ο εξωτερικός έλεγχος όμως ελέγχει μεταξύ άλλων αν ο εσωτερικός έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εσωτερικός έλεγχος των διαφόρων πολιτικών ομάδων και πολιτικών κομμάτων αν λοιπόν ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί σωστά, ιδεοδός προληπτικά, εντοπίζοντας, ανοιχνεύοντας και τακτοποιώντας τα του οίκου του οργανισμού χωρίς να χρειάζεται έτσι η παρέμβαση του εξωτερικού ελεγκτή. Αν ο εξωτερικός ελεγκτής ε, δει παρατυπίες δεν μπορεί παρά να τις αναφέρει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει ε, μια ε, διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Και αυτό αφορά και την παρέμβαση του κυρίου Χέφνερ. Εν παρόδο θα ήθελα να πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο ήδη έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την μεταφορά κάποιου ποσοστού των ε, πλεονασμάτων στον επόμενο χρόνο. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο πιστεύει ότι δεν είναι ε, τελεσίδικα λιμένο το θέμα αυτό της τήσιας μεταφοράς όπως αναφέρεται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να συζητείται μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αρχών του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, το θέμα της γραφειοκρατίας που ανέφερε ο κύριος ε, Χέφνερ. Δεν ε, αναμένει το ελεκτικό συνέδριο κάποιες προβλέψεις εξάμηνες για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε θεσπίσει δικούς σας κανόνες Γι' αυτό το ελεγκτικό συνέδριο συνεχώς απευθύνει κλήσεις στα θεσμικά όργανα, σε όλες τις αρχές, τις νομοθετικές, να εξυγχρονίσει τους κανονισμούς για να αποφεύγει ε, σύνθετα προβλήματα. Αυτού του τύπου η γραφειοκρατία δεν έχει σχεδιαστεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Αν υπάρχει, τότε υπάρχει νομοθεσία αν ε, υπάρξει θέμα κανονικότητας, ε, νομιμότητας, ε, εκεί υπάρχουν κανόνες, δεν έχουμε εμεί περιθώρια λιγμών. Τώρα, αυτό που είπατε για το μαντίο των δελφών το καταλαβαίνω, αλλά πολύ συχνά εμείς θα πρέπει να ε, τηρούμε κάποια ορολογία η οποία έχει αποφασιστεί από τα διεθνή λογιστικά ή ελεγκτικά πρότυπα. Πάμε τώρα στην, στην, στην τοποθέτηση της οργάνωσης διεθνής διαφάνεια. Παρακαλώ μην ξεπεράσετε το τέταρτο, γιατί πρέπει να έχουμε και άλλες τοποθετήσεις με τα κυρία Μίτερ Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον που έχετε για τις παρατηρήσεις και συστάσεις της Transparency International που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση ε, κατά της διαφθοράς. Γιατί μιλάμε σήμερα εδώ, γιατί η διεθνής διαφάνεια θεωρεί τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ως ε, περιοχή υψηλού κινδύνου διαφθοράς. Γι' αυτό είμαστε εδώ έχουμε εντοπίσει δύο τομείς ε, διαφθοράς στη χρηματοδότηση των κομμάτων. Πρώτον, ε, κατάχρηση των, του δημοσίου χρήματος για να παραμείνει κανείς στην εξουσία ή για ίδιο όφελος και αθέμητες επιρροές από κρυφές χορηγίες. Όταν δούμε αυτόν τον τομέα, δηλαδή διαφθορά στη χρηματοδότηση των κομμάτων, βλέπουμε δύο πηγές ή πρότυπα που πρέπει να τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα το ανέφερε ο κύριος Γκαλέα, είναι η Γκρέκο, στο Συμβούλιο της, ε, και ο κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. Και στο άρθρο 7, παράγραφος 3, αναφέρει σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βεβαίως έχει ε, και επικυρώσει τη σύμβαση αυτή κατά της διαφοράς, καθ' αυτή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μόνο τα 27 κρατη η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν υποχρεούται να βελτιώνει τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση υποψηφιωτήτων για ερετά δημόσια αξιώματα και να διασφαλίζει διαφάνεια στη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων. Η Διεθνής Διαφάνεια και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα ως οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών παρακολουθεί τις ιστοσελίδες ε, και τα έγγραφα που είναι ε, προσπελάσιμα στην κοινή γνώμη για να διαμορφώσει το βαθμό διαφάνειας από, μέσα από το πρίσμα εξωτερικού παρατηρητή με χρηματοδότηση. Ε, ο συνάδελφος ε, έχει επίση αναλύσει τα έγγραφα αυτά και είναι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Είδαμε λοιπόν τα δημόσια έγγραφα, αναλύσαμε και παρατηρήσαμε θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό που ε, αφιερώνεται στα πολιτικά κόμματα και που αυξάνει ετησίως κατά 25%, ενώ η συνολική αύξηση του προπολογισμού είναι πολύ πολύ μικρότερη και σημαντικά τμήματα του προϋπολογισμού διοχετεύονται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Επί τη βάση της ανάλυσης μας καταρτήσαμε ένα έγγραφο το οποίο μπορείτε στην είσοδο να το δείτε και υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Και εδώ έχουμε πέντε κύριες παρατηρήσεις που συνοψίζουμε εδώ. Καταρχήν, είναι καλό ότι οι εκθέσεις από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα είναι online, επιγραμμικά, αυτό είναι καλό. Επίσης εκτιμούμε το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις εκθέσεις είναι τυποποιημένες και χρησιμοποιούν τυποποιημένο πίνακα που έχει προταθεί από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης χαιρόμεθα διότι οι εκθέσεις έχουν ελεγχθεί. Όμως, και πάμε τώρα στην δεύτερη παρατήρηση, το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επισήμανε λήψεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο δηλαδή επισήμανε τις ε, λήψεις στην διαφάνεια της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών κομμάτων κατά τη διαδικασία απαλλαγής του προϋπολογισμού του 2008. Και σε αυτή την κριτική επίκριση αναφέρεται ότι οι εκθέσεις αναφέρονται μόνο ως ε, έγγραφα του προσχεδίου του προϋπολογισμού που έχει σκαναριστεί και ότι δεν υπάρχει τυποποιημένη δυνατότητα ε, σύγκρισης ε, που να διευκολύνει εμάς που βλέπουμε ως εξωτερική τη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να κατεβάσουμε σε μορφή Excel τα δεδομένα και να κάνουμε σύγκριση. Ενώ αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Η διαθεσιμότητα των εγγράφων για ανάλυση δεν παρέχεται δηλαδή εκείνη τη χρονική στιγμή. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι στην τυποποιημένη μορφή που υπάρχει, που παρέχεται, αναφέρονται εισφορές σε είδος, αλλά όχι χορηγίες σε είδος. Που αυτό το τελευταίο πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Και μόνο δύο κόμματα αναφέρουν ότι έλαβαν χορηγίες το 2009. Δεν το αναφέρουν όλα. Επίσης, ανησυχούμε διότι δεν υπάρχει με συνέπεια υποβολή εκθέσεων για τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας του 2009 και λείπουν οι λεπτομέρειες για τα ε, έσοδα-έξοδα δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία. Υπάρχει και σχετική έλλειψη διατάξεων που να αφορούν αυτό το θέμα στον παρόντα κανονισμό. Θα θέλαμε πάρα πολύ αν την ε, επόμενη περίοδο η κοινωνία των πολιτών που υποτίθεται ότι παρακολουθεί τη χρηματοδότηση μπορούσε ε, να διευκολυνθεί και να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις μας. Αυτό που θέλει η κοινωνία των πολιτών είναι πλήρης και 100% τυποποιημένες εκθέσεις από όλα τα πολιτικά κόμματα. Οι εκθέσεις θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμες και συγκρίσιμες online, συμπεριλαμβάνοντας μορφότυπους που επιτρέπουν ανοιχτή προσθήκη δεδομένων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις χορηγίες περιλαμβάνοντας και σε είδος υποστήριξη για εκδηλώσεις κομμάτων, για παράδειγμα, και θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά αποθέματα, όπως είπε και ο κύριος Γκαλέα. Και τέλος, μια πολύ σημαντική σύσταση θα πρέπει να είναι η εξής. Εν ώψη των εκλογών το 2014, η Transparency International θα ήθελε ε, μια ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρηματοδότηση των εκλογών, όπως είπε και ο κύριος Γκαλέα. Αυτό θεωρητικά θα πρέπει να γίνεται και να συνοδεύεται και μια αξιολόγηση του κινδύνου. Τέλος, πολύ σημαντικό, συμφωνούμε με την πρόταση του κυρίου Γκαλέα για αυξημένα μέτρα ελέγχου που χρειάζονται για να προστατεύονται τα δημοσιονομικά της Ένωσης σε τελευταία ανάλυση και συμφωνούμε και με την πρόταση του κυρίου Μόρλοκ νωρίτερα για τη ζωτική σημασία των ε, κυρώσεων για την προστασία των, των ενωσιακών κονδυλίων και για ε, την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων αν σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα διαπιστωθεί διασπάθηση κονδυλίων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το περιεχόμενο, τη συντομία και τα έγγραφα που μας στείλατε. Ο κύριος Νταφ. Um, uh, Καταρχήν δεν θα πρέπει να μεγεθύνουμε, να διωγγώνουμε τα προβλήματα. Και η ιδέα ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα διαφύρονται από την άσκηση εξουσίας ε, είναι παράλογη η αιτία του κακού, η αιτία του προβλήματος είναι ένας αλλοπρόσαλος δημοσιονομικός κανονισμός, ένας τελείως παρανοϊκός δημοσιονομικός κανονισμός για την υποστήριξη των κομμάτων που απαγορεύει από τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενεργούν ως πολιτικά κόμματα ουσιαστικά. Τους απαγορεύει δηλαδή τη διεξαγωγή εκστρατεία. Τους απαγορεύει να υποστηρίζουν υποψηφίους, συγκεκριμένους υποψηφίους και όχι μόνο απαγορεύει την άμεση υποστήριξη εθνικών πολιτικών κομμάτων, αλλά και την έμεση υποστήριξη απαγορεύει. Όλα αυτά είναι παράλογα, είναι φως φανάρι. Κάτι τέτοιο οδηγεί και μάλιστα υποχρεώνει τα κόμματα να προσφύγουν σε φάνταστη λογιστική και να εφαρμόζουν αυτή τη δημιουργική λογιστική προκειμένου να αλλοιώνουν τα στατιστικά στοιχεία και τα λογιστικά του στοιχεία. Ελπίζω, η κυρία Γιαννάκου, να διαγράψει πλήρως το άρθρο 7 του δημοσιονομικού κανονισμού και να επιτρέψει τα Πράγματα που σήμερα απαγορεύονται, γιατί είναι αδιανόητο να προσβλέπουμε σε πανευρωπαϊκή εκλογική λίστα και να απαγορεύουμε την ε, διεξαγωγή εξτρατείας. Δεν μπορούμε να απαγορεύουμε και τη χρηματοδότηση τέτοιων εξτρατείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τίποτα άλλο να μην κάνουμε στο νομικό καθεστώ, στην αλλαγή του νομικού καθεστώτο ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων μέχρι το 2014, θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να το κάνουμε, αυτή τη διαγραφή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντεμπούτ, ο οποίος είναι και ο γραμματέας του ε- Ευρωπαϊκού ΕΛΚ, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να δώσουμε τη γνώμη μας για την ε, αναθεώρηση ε, που προτείνεται και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την Επιτροπή για την πρωτοβουλία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμβολή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη συμβολή των ειδικών από τα πανεπιστήμια, από το ελεγκτικό συνέδριο, πολύ χρήσιμα όλα αυτά, και δείχνουν ότι υπάρχει ευρεία συνένεση. Ε, τα ευρωπαϊκά κόμματα είναι σχετικά ε, καινούρια, ε, ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 70 και του 80, χρειάστηκε όμως μια γενεά μέχρι, περάσουν 25 χρόνια περίπου μέχρι να θεσμοθετηθούμε στις συνθήκες. Ακόμα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, είναι μακρύς ο δρόμος. Ε, σε αυτή τη σειρά που εκπροσωπούνται τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αναφέρεται το Group PPE, Group SD, Group ALDE. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσουμε ε, μάχη για την ταυτότητά μας. Δεν είμαστε εμείς προσαρτήματα των κομμάτων, είμαστε ανεξάρτητα πολιτικά κόμματα. Κάναμε πολύ δρόμο από το Μάστρι στη Νίκαια, του κανονισμό του 2004, την αναθεώρηση και τώρα έχουμε μια εξαιρετική αναθεώρηση των προηγουμένων κανονισμών με πολλά μέτρα που θα διευκολύνουν τη ζωή μας, που θα ε, μειώσουν γραφειοκρατίες ε, και διοικητικά ε, βάρη Επίσης είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπε η Transparency International. Όμως ε, μην περιμένετε να έχουμε ε, φάκελο Excel με τα δεδομένα μας ε, επιγραμμικά online. Αυτό δεν το κάνουν τα κόμματα. Υπάρχει στο προσχέδιο του προπολογισμού, στοιχεία για τον προπολογισμό, αλλά Excel file δεν μπορεί ποτέ να περάσει στο διαδίκτυο. Κατά τα άλλα είμαστε υπέρ των εκ των ελέγχων, ε, των... Ε, επίσης για τους ε, ελεγκτές υπάρχει πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινό εξωτερικός ελεγκτής που θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία, εφόσον θα έχουμε ευρωπαϊκό καθεστώς, γιατί τώρα είμαστε ε, λειτουργούμε βάσει του βελγικού νόμου για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και η νομοθεσία αυτή προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ορισμός ελεγκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο για να ανταποκριθούμε στα θεμητά σα ερωτήματα και αιτήματα. Και μια και μιλάμε και για, τον, για το καταστατικό, μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι χαιρόμεθα που καταφέραμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, πέρα από το 2004 και το 2007. Μιλάμε για την πολιτική, μας, πολιτική σημασία στην πανευρωπαϊκή αυτή συζήτηση, η οποία βέβαια θα ε, πρέπει να στηρίζεται στην νομική και οικονομική ε, νομιμότητα. Ε, αυτά που είπε ο κ. Σέφνη το πρωί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί μη διαφοροποιούμε μεταξύ αναγνώρισης πολιτικού κόμματος και σε δεύτερο ε, βήμα θα πρέπει να οριστούν κριτήρια για τη χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ σημαντικό για την εσωτερική εσωκομματική δημοκρατία. Ναι, Όλοι μας έχουμε καταστατικά, αλλά προφανώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ισοκομματική δημοκρατία με online ερωτηματολόγια κλπ. Το, η ατομική ιδιότητα του μέλους, ναι, αλλά με μεγάλη προσοχή. Και οι σοσιαλιστές και άλλοι έχουν σύστημα ε, οπαδών, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Έχουν δικαίωμα να λάβουν το λόγο, αλλά όχι να ψηφίζουν. Θα πρέπει να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ. Είμαστε μια συμμαχία κομμάτων μελών και τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα ίσως υβριδική μορφή ε, όπου θα έχουμε τα κόμματα και μονομενά δικαιώματα. Και εκεί το δικαίωμα ψήφου είναι πολύ σημαντικό. Πάντως υπάρχει αυτή, αυτό, αυτή η δυναμική που θα μας κάνει σημαντικούς παράγοντες ε, διεθνώς. Υπάρχει και η ε, έκθεση του κυρίου Άντριου Ντάφ για την εκλογή ε, αριθμού ε, ευρωβουλευτών, 25, 50, 10, δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός, είναι συμβολικό. Μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε τη συνείδηση των ψηφοφόρων των εκλογέων σε ευρωεκλογές. Και το 2004 προσπαθήσαμε και μία από τις παρεμβάσεις μας δίνει την νομιμότητα να είμαστε γνήσιοι παράγοντες. Υπάρχει και η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Μην υποτιμούμε το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα πολιτικά κόμματα εδώ. Ε, σας ευχαριστώ, εκφράζω εδώ ε, όλο το, το κόμμα μου. Ε, ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα θέματά μας και ευχαριστούμε πολύ και για την υποστήριξη που μας παρήχατε. Ευχαριστώ. Ευχ, σας ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο στην κυρία Γιαννάκου για το συμπέρασμα. Κύριε Πρόεδρε, η ακρόαση αυτή πραγματικά υπήρξε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Συμπληρούμενη από τους δύο τελευταίους ομιλητές, τον καθηγητή κύριο Γκαλέα του Ελεκτικού Συνεδρίου και την κυρία Φιτμάγια από την Διεθνή Διαφάνεια, πραγματικά αναδεικνύονται όλα τα ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δημιουργία ε, στάτους για τα ευρωπαϊκά κόμματα μάλλον τα κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως πολύ σωστά τόνισε ο κύριος Γκαλέα, διότι έτσι γράφει η συνθήκη. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που ζητούμε για το στάτους των ευρωπαϊκών κομμάτων, δηλαδή να υπάρχει μία πολιτική, νομική και φορολογική προσωπικότητα που θα αφορά τα κόμματα και το στάφ και το σημειώνω αυτό διότι του Γενικού Γραμματέως το σημείωμα λέει ότι αυτό το τελευταίο, το φορολογικό δεν είναι δυνατόν, ε, ασφαλώς δεν ζητείται να δοθεί στα staff των πολιτικών κομμάτων στάτους των ε, υπαλλήλων οι οποίοι έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό. Αλλά σας θυμίζω ότι υπάρχει στάτους για τους συνεργάτες των βουλευτών που δεν επιλέγονται με διαγωνισμό και υπάρχει και στάτους για ένα πλήθος συμβασιούχων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά όργανα που δεν προσλαμβάνονται με διαγωνισμό. Σας θυμίζω ότι η Κομισιόν έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 6.000 αζάν ταμπορέ. Επομένως δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα εκεί για οποιαδήποτε εξομοίωση. Το θέμα είναι θα έχουμε νομική προσωπικότητα και πραγματικό στάτους για όλους. Το ερώτημα που προέκυψε από τη Διεθνή Διαφάνεια και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου είναι μήπως γίνεται κατάχρηση εξουσίας από ε, το γεγονός ότι διαχειρίζονται χρήματα. Όμως, όπως εμείς βλέπουμε το βήμα το επόμενο που θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή τα κόμματα αυτά να έχουν τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορούν να υπάρχουν οπαδοί ή και μέλη αυτοί που θέλουν να γίνουν κατευθείαν μέλη. Με κάποιο ρόλο φυσικά ο οποίος θα είναι διαφορετικός από τα κόμματα μέλη που απαρτίζουν ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Δεν νομίζω ότι επιτρέπει να κάνουμε σκέψεις για κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά. Άλλωστε το Ελληνικό συνέδριο είναι πολύ αυστηρό στις κρίσεις του για τα ζητήματα αυτά. Και βεβαίως τίποτα δεν το εμποδίζει να κάνει και ένα είδος προληπτικού ελέγχου και να προειδοποιεί ε, τους θεσμούς αυτούς για το πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους. Επομένως νομίζω ότι έχουμε τους μηχανισμούς ε, οι οποίοι μπορούν να μας προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους παρέστησαν σήμερα εδώ. Τους καθηγητές Πανεπιστημίου, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου, την εκπρόσωπο της Διεθνούς Διαφάνειας, αλλά κυρίως ε, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συζήτηση που έγινε το πρωί με την παρουσία όλων προέδρων ή γενικών γραμματέων ε, ή υπευθύνων αξιωματούχων των διαφόρων πολιτικών κομμάτων και σχηματισμών που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν πολιτικό ρόλο στο επίπεδο της Ευρώπης μέσω των εθνικών κομμάτων που είναι μέλη τους αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή εκτός από την παρακολούθηση της χρηματοδότησής τους και τις όποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμε εκεί, να δώσουμε στα κόμματα αυτά την ευκαιρία να έχουν ένα νομικό καθεστώς το οποίο θα είναι σεβαστό σε όλα τα κράτη-μέλη. Διότι αν θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά, αυτή τη στιγμή το νομικό καθεστώς που ισχύει για διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση στο Βέλγιο μπορεί κάλλιστα να μην είναι σεβαστό ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ισπανία, ούτε πουθενά άλλου. Άρα μας χρειάζεται ένα καθεστώς που δεν θα έρχεται σε σύγκρουση με τα συντάγματα των κρατών μελών και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε αυτό το οποίο θα έχει πολιτικό βάρος, νομική ισχύ και φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι σεβαστό για όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι μπορούμε κάλλιστα να έρθουμε στο ζήτημα που περιλαμβάνει η έκθεση του κυρίου Νταφ για το πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία λίστα καταρχήν με έναν αριθμό τον οποίο μπορούμε να το βρούμε. Μπορεί να είναι 25, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 15, σημασία έχει η αρχή. Τότε μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για να έχουμε μια τέτοια λίστα. Δεν πιστεύω όμως ότι μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα χωρίς να έχουμε ένα στάτους ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων γιατί μπορεί να προκύψουν διάφορα ζητήματα που θα οφείλονται στις διαφορετικές νομοθεσίες στα κράτη-μέλη και στις διαφορετικές συνταγματικές ρυθμίσεις και να μας φέρουν μπροστά σε αδιέξοδα και σε σοβαρά προβλήματα. Κύριε Πρόεδρε, όλα όσα ελέγχθησαν είναι πολύτιμα για την έκθεση η οποία θα συνταχθεί. Πιστεύω ότι όλοι κατέληξαν πάντως σε ένα συμπέρασμα. Ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα πραγματικό στάτους σεβαστό από όλε τις πλευρές. Λεπτομέρειες που θα αφορούν, αν ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα θα είναι μέλη, πώ θα ρυθμίζονται οι σχέσει με τα κόμματα κτλ. Αυτές μπορούμε να τις βρούμε. Σημασία έχει ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Φυσικά συντάσσοντας μία έκθεση η οποία θα αποτιμά με βάση την έκθεση του Γενικού Γραμματέα η οποία είναι πολύ καλή ε, θα αποτιμά τη χρηματοδότηση αν ο σκοπός της επετεύχθη και αν πραγματικά τα πράγματα είναι διαφανή και σωστά. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τελικά όλα τα μέλη της Επιτροπής και τους συνεργάτες που συμμετείχαν εδώ σήμερα σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση που νομίζω ότι ε, μας ε, κίνησε το ενδιαφέρον και δεν άφησε κανέναν μας να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Eh. Σας ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου και σας ευχαριστώ και προκαταβολικά για το μέλλον διότι στις 31 έχουμε την έκθεσή σας. Δεν ξέρω εάν λαμβάνοντας υπόψη όλο αυτό το πλουσιότατο υλικό που συλλέξαμε σήμερα θα καταφέρετε να επεξεργαστείτε, να τα εντάξετε όλα αυτά και να επεξεργαστείτε την έκθεση. Λοιπόν, η επόμενη συνεδρίαση θα είναι τη Δευτέρα στις 31 Φεβρουαρίου και θα έχουμε μετά και την 1η Φεβρουαρίου και 7 Φεβρουαρίου θα έχουμε μια άλλη συνεδρίαση έκτακτη για την έκθεση ΝΤΑΦΑ σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πέρα συνεδρία συνεδρίες